Chers collègues, je propose de commencer notre réunion. Ας ξεκινήσουμε. Καλημέρα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να επισημάνω δύο τραγουδίσεις της ημέρας διάταξης. Η πρώτη φορά το σημείο 21 και την ψηφοφορία του συναδέλφου Σαρικάς που θα μετατεθεί ως τελευταία μετά το σημείο 30. Στο σημείο 16, δηλαδή σε τη φορά της ε, διαπραγματεύση. για την ενδοπιχειρησιακή μετάθεση, θα το εξετάσουμε ως πρώτο σημείο μετά τις ψηφοφορίες. Υπάρχουν αντιρρήσεις? Όχι προτείνω λοιπόν να περάσουμε το σημείο 17 όπου πρέπει να σας ε, παρουσιάσω τις συμβαστικές τροπολογίες που κατατέθηκαν ε, επί της ε, γνωμοδότησης που εκπονούμε και εκπονεί η Επιτροπή Προπολογισμού με τον απολογισμό των διαπραγματεύσεων για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ήδη έχουμε συζητήσει αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης και υπήρξε σημαντικός αριθμός ε, τροπολογιών. Οι περισσότερες είχαν κατατεθεί από τους συναδέλφους Χάρκιν και Λάμπερτ. Επί της ουσίας ε, μπορώ να συμφωνήσω με αυτές τις τροπολογίες. Οι δύο συμβαστικές τροπολογίες που σας ε, πρότεινα αφορούν ε, την τροπολογία 2 του Τζιν Λάμπερτ, δική μου 3 και την τροπολογία 4 της κυρίας Χάρκιν. που αφορούν ε, τις συνθήκες υπό τις οποίες ε, συλλέγονται τα δεδομένα ε, της απασχόλησης. Είναι μια τροπολογία που συνθέτει διαφορετικές απόψεις και δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Στην Β συνθέτουμε τις τροπολογίες 13, 14 και 15 Θέλουμε να βελτιώσουμε τον τρόπο διαπραγμάτευσης ε, των οριζόντων ε, θεμάτων. και να εξετάσουμε πλανεκτήματα ε, της έκθεσης ε, EASY και να καταδείξουμε πως αυτές οι διαπραγματεύσεις κάποιες φορές αντιμετώπισαν δυσκολίες ε, εξαιτία αυτής της κατάστασης. des autres amendements. Για τις υπόλοιπες τροπολογίες είμαι υπέρ. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε να περάσουμε σε ψήφιση αυτής της νομοδότησης που θα ενισχύσει ε, τη φωνή της Επιτροπής μας, αλλά και της Επιτροπής Ευρωπολογισμών. Έγιναν παρατηρήσεις και στη διάσκεψη των Προέδρων για αυτή την ε, έκθεση και επειδή υπάρχει και μια παράλληλη έκθεση που συζητείται στην ε, Επιτροπή ΑΦΚΟ, θα συζητήσω με του συναδέλφους ε, που την έχουν αναλάβει που θα εξετάσουν σε βάθος την ουσία αυτής της έκθεσης στην Επιτροπή Προπολογισμών γιατί εκεί αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι ότι σε αυτή την επιτροπή, στη δική τους, θα πρέπει να εξετάσουν μόνο τα ζητήματα που ε, αφορούν τις διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και ε, τα ζητήματα σταματικών υποθέσεων θα πρέπει να τα εξετάσουμε στο ιστορικό του Κοινοβουλίου. Εγώ διαφωνώ με αυτό το στοιχείο, γι' αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε αυτές τις δύο τροπολογίες που ε, διευκρινίζουν τη δική μας προσέγγιση ως προς αυτές τις διαπραγματεύσεις. Οι συνάδελφοι που κατέθεσαν τις τροπολογίες θέλουν ε, να παρέμβουν και πάλι. Υπάρχουν ε, αντιρρήσεις ε, στις συμβαστικές τροπολογίες. Όχι. Όλα καλά λοιπόν. Μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο σημείο της μέσης διάταξης. Να δώσω το λόγο στην κυρία Σοβιέτσκα. για να μας ενημερώσει για τον έκτο και 7ο τριμερή διάλογο που έλαβε χώρα προχθές στο πλαίσιο της ε, διαπραγματεύσης ε, για την εφαρμογή της οδηγίας απόσπασης εργαζομένων. Πριν σας δώσω το λόγο όμως, θα ήθελα να πω το εξή. Ακούγονται φήμες ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις παίρνουν πολύ χρόνο. Πρέπει να πω ότι αυτό δεν ευσταθεί. Οποιοςδήποτε έχει συμμετάσχει σε τριμερείς διαλόγους, σε ένα νομοθετικό κείμενο, γνωρίζει ότι είναι μια χρονοβρό διαδικασία. Υπερθυμίζω ότι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τα Ευρωπαϊκά Κοινωνικά Ταμεία, που αφορούσε ποια άρθρα, το 19, 30 άρθρα περίπου, 30 άρθρα. Διεξήγαμε πάνω από 30 τριμερείς διαλόγους. Και εδώ βρισκόμαστε μόλις στον 7ο. Και ήδη έχουμε εξετάσει όλα τα ακαθόδη ζητήματα. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουν εδώ αυτές οι φήμες ότι υποτίθεται αυτές οι πραγματεύσεις ε, παίρνουν πολύ χρόνο. Δεν ισχύει οι θέσει Κοινοβουλίου και Συμβουλίου διαφέρουν. Είναι λογικό λοιπόν να χρειαζόμαστε ένα διάστημα για να παραθέσουμε ξεκάθαρα τις ε, θέσεις μας ε, στο Συμβούλιο. Προκειμένου να ακούσουν και αυτοί τις δικές μας απόψεις. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο για την ε, την συνάδελφη συγγήτρια για την επιμονή της. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλη την ομάδα και να αναφέρω και να επαληθεύσω τα όσα είπατε και εσείς μόλις τώρα. Γιατί πράγματι γίνονται ταχύτατα οι διαπραγματεύσεις. Προφανώς δεν είναι εύκολες και γι' αυτό πρέπει να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο και θα ήθελα να παρουσιάσω την κατάσταση όσα έχει αυτή τη στιγμή. Μετά τις ε, τελευταίες συνεδριάσεις της Επιτροπής, όπου έδωσα έκθεση για την, Επιτροπή, την οδηγία ε, εφαρμογής της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων, είχαμε συνεδριάσεις στις 6 και στις 11 Φεβρουαρίου. Είχαμε συζητήσει για το άρθρο 9 που που είχε προετοιμάσει το Συμβούλιο και συμβαστικές ε, προτάσεις ε, οδήγησαν σε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η Επιτροπή ήθελε ανοιχτό κατάλογο ελέγχων και επιθεωρήσεων και δεν ήθελαν τίποτα επιπρόσθετο που πρότεινε το Συμβούλιο. Ακόμα και αν αυτά τα μέτρα ήταν ε, ανάλογα και κατά των διακρίσεων. Ε, άλλη σημεία συζήτηση ήταν και η διατήρηση των δεδομένων και των εγγράφων που πρέπει να είναι υποχρεωτική σε όλα τα κρατημέλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε να στείλει στην Επιτροπή πληροφορίε για επιπλέον ε, μέτρα ελέγχου, αλλά υπόθηκε ότι δεν συμφωνούν όλοι με τις υποχρεωτικέ κοινοποιήσει. Η Προεδρία, προκειμένου να υπάρξει συμβασμός ε, με το Κοινοβούλιο, θα το εξετάσουμε από κοινού στις 18 Φεβρουαρίου. Και στον τελευταίο τριμερή διάλογο εξετάσαμε το άρθρο 12 για την ε, ε, νομική ευθύνη. Ε, το Κοινοβούλιο έχει πολύ συγκεκριμένη θέση και βάσει των όσων έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή Απασχόλησης δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τέτοιο μηχανισμό σε όλους τους κλάδους, σε όλη την ε, αλυσίδα. Θα γίνει λοιπόν μια ανταλλαγή απόψεων, θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση από την Επιτροπή για τους ε, μηχανισμούς ε, νομικής υπετιότητα που υπάρχουν στα άλλα κράτη-μέλη. Η Προεδρία θα παρουσιάσει συμβαστική πρόταση την Παρασκευή και θα εξεταστεί στον επόμενο τριμερ διάλογο. Στην τελευταία συνεδρίαση τριμερούς διαλόγου ολοκληρώσαμε τις συζητήσεις για τα άρθρα 6, 7, 8 και 11. Εδώ στο 6 η Ελληνική Προεδρία εισήγαγε μια προθεσμία 20 ημερών αντί για 25 και μιλά... Περνάμε στο 27, στο 7, συγγνώμη, για τον κύριο ρόλο της ε, χώρας ε, που, από την οποία φεύγουν οι εργαζόμενοι. Αρχικά έγινε δεκτή η πρόταση του Κοινοβουλίου για τη συνεργασία μεταξύ των μελών μεταξύ των δύο χωρών προέλευσης και υποδοχής. Στο 8 η Προεδρία συμφώνησε να στηρίξουμε την πρωτοβουλία για να υπάρξει μια διάδοση πληροφοριών προς ε, τους αποσπασμένους εργαζομένους και εργάτες. Το άρθρο 10 για τις επιθεωρήσεις συμφωνήσαν ε, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο ότι τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση να διεξαγάγουν αποτελεσματικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις θα πρέπει να υπάρξει και η μεξολόγηση κινδύνου που είναι το καλύτερο μέσο, όμως τα κράτη-μέλη θα επιλέξουν ε, τον ε, τρόπο που επιθυμούν. Άρθρο 11. Με υποχρέωση τα κράτη-μέλη εισαγωγή ενός μηχανισμού που επιτρέπουν ε, τα, εργαζομένους ε, να απολάβουν των δικαιωμάτων τους, των εργοδοτών. Βεβαίως συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα επιδόματα αλλά και τις ε, φορολογικές υποχρεώσεις ε, που τους αναλογούν. Στο IMI τώρα, στο 18, αποφασίστηκε, μάλλον το, το Συμβούλιο θεωρεί ότι πρέπει να αποτελεί υποχρεωτικό μηχανισμό και τα κάτι μελη θεωρούν ότι θα πρέπει να πρόκειται για διμερή συμφωνία. Θα υπάρξει ακόμα τριμερή διάλογο για το κεφάλαιο 6, διασυνοριακή επιβολή προστήμων και τελών. Και θα γίνει και άλλο τριμερή διάλογο 18, 19 και 20 Φεβρουαρίου και ελπίζουμε εκεί να εξετάσουμε τα άρθρα 9 και 12 και μέχρι τα τέλη του μήνα να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Θα ήθελε κάποιος να παρεμβεί. Τα άλλα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ίσως ο Στίβεν Χιούζ, όχι φαίνεται ότι δεν έχει κάτι να προσθέσει. Κάποιος άλλος ή διασαφήσεις, θέλετε κάτι. Εγώ απλώς θα ήθελα να προσθέσω ένα στοιχείο. Καταρχήν ε, ευχαριστούμε την εισηγήτρια για αυτή την πιστή ε, αναμετάδοση και σε ε, σχέση με το πρώτο σκέλος μπορούμε να λάβουμε υπόψη την προστασία των εργαζομένων μέσα σε αυτό το πλαίσιο έτσι ώστε να ευνοούνται κατά το δυνατόν και να πω ότι στην πρωτοβουλία μας γνωρίζουμε ότι το κείμενο βρήθη από ρήτρες αναθεώρησης. Το ξέρουμε αυτό. Όταν η διαπραγμάτευση είναι δύσκολη, ε, τότε θέλουμε οπωσδήποτε να φτάσουμε σε μια συμφωνία και λέμε ωραία θα αναθεωρήσουμε όποτε μπορέσουμε και ε, προσθέτουμε ένα άρθρο, μια ρήτρα αναθεώρησης. Άρα το ε, κείμενο βρίθει από ρήτρες αναθεώρησης σε όλα τα άρθρα ε, όπου ανακύπτουν και ζητήματα χρονισμού παράλογα. Δηλαδή η οδηγία χρειάζεται δύο χρόνια, χρόνια για να τεθεί σε ισχύ. Η Επιτροπή θα προβεί σε μια έκθεση αξιολόγησης μετά από πέντε χρόνια και θα έχουμε την αναθεώρηση μετά από τρία χρόνια. Δηλαδή θα αναθεωρήσουμε την οδηγία πριν αποφανθεί η Επιτροπή με έκθεση αξιολόγησης. Ως καλοί νομοθέτες λοιπόν είπαμε ότι τα πράγματα δεν έχουν καλώς. Άρα είτε η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να ε, αλλάξουν θέση και μας είπαν ε, ότι έχουμε δίκιο. έτσι ώστε να αναθέσουμε εντολή στην Επιτροπή για να βρει μία οριζόντια λύση, μία οριζόντια ρήτρα, περιλαμβάνοντας το άρθρο 9 που για μας είναι πολύ σημαντικό. Αυτό ήθελα να υπενθυμίσω και δεύτερον, σε σχέση με το τελευταίο σημείο που έθιξε η εισηγήτρια, το άρθρο 18 που θέτει σε εφαρμογή ένα σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά έτσι ώστε η Επιτροπή να συλλέξει τις πληροφορίες σε σχέση με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το σύστημα αυτό ε, δεν έχει προσαρμοστεί για τις ανταλλαγές απόψεων που αφορούν τους αποσπασμένους εργαζόμενους μέσα στα πλαίσια των μητρών όπου έχουν ε, εγγραφεί οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι. Άρα η Επιτροπή διαχρονικά θα πρέπει να ασχοληθεί ε, με αυτό το ζήτημα. Υπάρχει κάτι άλλο το ενδιαφέρον που αγνούσε η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης όταν η Κομισιόν έχει πληροφορίες για τους αποσπασμένους τις έχει μέσα από τα δελτία Α1. Γι' αυτό είναι ύψη της σημασίας για εμάς σε αυτά τα δελτία Α1 να υπάρχει ειδική μνήμα για το θέμα που μας απασχολεί. δηλαδή τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένα μέσα πληροφόρησης για το τι ισχύει για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο της συζήτησης. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο όχι, όπως είπε και η συγγήτρια, σήμερα το απόγευμα θα γίνει η επόμενη ανταλλαγή απόψεων με ένα χρονοδιάγραμμα πολύ πιεσμένο, συνεργασία με το Συμβούλιο και την Κομισιόν και είχαμε και τριμερή διάλογο προχτές. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να αρκεστούμε σε αυτό το χρονοδιάγραμμα με ανταλλαγές απόψεων στην Κορεπέρ την Παρασκευή και την επόμενη Τετάρτη. Άρα η ομάδα διαπραγμάτευσης θέλει να φτάσει σε αίσιο πέρας και ελπίζω να πραγματοποιηθεί αυτό. Πολλά εξαρτώνται από τι θα γίνει σήμερα το απόγευμα. Αλλά δεν έχουμε δύσκολα άρθρα για σήμερα το απόγευμα. Θα τα διατρέξουμε Άρα θα δούμε τι θα γίνει μεταξύ εκπροσώπων των κρατών μελών στην Κορεπέρ την Παρασκευή και την εντολή που θα δώσουν τα κράτη-μέλη με βάση τις συζητήσεις που έγιναν το Δεκέμβριο. Νομίζω ότι έχετε όλα τα στοιχεία για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων που ελπίζω να μας κινητοποιήσει όλους πέρα από την ομάδα διαπραγμάτευσης καθεαυτή. Φτάνουμε τώρα στην ώρα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Έχετε τις κάρτες σας. Εγώ έχω τη δική μου, εσείς. Oui, tout le monde a sa Έχετε όλες τις κάρτες σας. Alors, euh, nous allons commencer. nous allons commencer au point 19. Θα αρχίσουμε με το σημείο 19. Τα αποτελέσματα της συνεργασίας με το Συμβούλιο για την ενισχυμένη συνεργασία των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης. Πρόκειται για τα αποτελέσματα της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου με ε, αίσιο πέρα στις 29 Ιανουαρίου 2014 και που επιβεβαιώθηκε από την Κορεπέρ της 7 Φεβρουαρίου 2014. Φρεντερίκ Ταρντέν είχε αναλάβει τις διαδικασίες. Αρχίζει η ψηφοφορία. Tout le monde a pu voter. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 28 υπέρ, 1 κατά, 3 αποχές η κοινή θέση εγκρίνεται. Να συγχαρούμε τον εισηγητή μας και όλη την ομάδα διαπραγμάτευσης. Ως προς σημείο 20 θα πρέπει να ψηφίσουμε για τη γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Προϋπολογισμού για την Κοινοτοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μέσα στα πλαίσια της κοινότητας της ε, Βαλένθια στον τομέα της ε, κλωστοεφαντουργίας στην Ισπανία. Πρόκειται για την κινητοποίηση του Ταμείου υπό το καθεστώς της ε, προηγούμενης διαφθέτησης. Υπέρ παρακαλώ της επιστολής. Α, όχι, με συγχωρείτε, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία 31 υπέρ, μία ψήφο κατά, καμία αποχή. Άρα η γνωμοδότηση είναι θετική και θα τη διαβιβάσουμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Φτάνουμε τώρα στην έναρξη των εργασιών μας, στο σημείο 22, όπου θα ψηφίσουμε την έκθεση Τσάμπα Όρη μέσα στα πλαίσια της, ε, της ε, τριμερούς κοινωνικής ε, συνόδου. Πριν ψηφίσουμε, ζητώ συγγνώμη γιατί χτες δεν ήμουν στην ψηφοφορία, αλλά θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια. Να σας πω ότι πρόκειται για μια ενδιάμεση έκθεση. Δεν είναι το τελικό πρόγραμμα, διότι δυνάμει της διαδικασίας του άρθρου 81 το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνενέσει, άρα πρόκειται για μια διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο πριν αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που θα ήθελα να και να σας υπενθυμίσω. Δεύτερον, επειδή πρόκειται για διαδικασία συνένεσης, συνενετική δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο το έθιξαν το θέμα οι συντονιστές και θα πρέπει να το διασαφίσουμε. Επίσημα δεν έχουμε λάβει τις προτάσεις του Συμβουλίου διότι το Συμβούλιο πρέπει να διαβολευτεί με τα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη έχουν μία προθεσμία για κινητοποίηση και για να ε, με τα εθνικά τους κοινοβούλια. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία δεν απάντησαν στην προθεσμία των τεσσάρων εβδομάδων δεν έχουν ακόμα αποφανθεί, άρα το Συμβούλιο δεν μπορεί να διαβιβάσει επίσημα τη θέση τους. Άρα δεν ξέρουμε πώς έχει η διαπραγμάτευση, πώς θα καταλήξει. Αυτό σημαίνει ότι όταν εξετάσαμε για πρώτη φορά την έκθεση Τσάμπα Ορί, ότι μας ελέγχθη από την Κομισιόν ήταν λανθασμένο διότι στόχος αυτής της ε, διαδικασίας ήταν να επιτρέψουμε επίσημα στον πρόεδρο Χέρμαν Rompuy να συνδράμει στις 20 Μαρτίου στη διάσκεψη, στην τριμερή διάσκεψη ε, κορυφής. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει δύναμη της ε, τρέχουσας νομοθεσίας. Επειδή πρέπει να ε, ζητήσουμε τη γνώμη των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων, η τροποποίηση της απόφασης δεν θα γίνει πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, του, το αιαρινό ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. θα πρέπει να σας εκφράσω και την απογοήτευσή μου δηλαδή ικανοποίηση και απογοήτευση στο συμβασμό Β. Ικανοποίηση γιατί βλέπω ότι ο ή διαδοχός μου θα εκπροσωπήσει το Κοινοβούλιο στον, στην τριμερή διάσκεψη κορυφής, αλλά νομίζω ότι έχουμε κατεβάσει τον πύχη. Δεν βλέπω γιατί το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι πάντα παρατηρητής σε αυτές τις ε, τριμερείς διασκέψεις. Εδώ προβλέπετε απλώς να ε, προσκαλείτε με βάση την ατζέντα που προβλέπετε. Εγώ θα πρότεινα λοιπόν ενδεχομένως την τελική ψηφοφορία επειδή δεν θα υπάρξει τελική διευθέτηση του ζητήματος ε, σε αυτή τη θητεία, να ζητήσουμε από την Ολομέλεια μία εντολή διαπραγματεύσεων για να δούμε κατά πόσο έχει βρεθεί η σωστή ισορροπία στο κείμενο που θα ψηφίσουμε σήμερα. Αυτά σας ε, προτείνω. Δεν ξέρω αν θέλει κάτι να μας πει ο εισηγητής. Φαίνεται πως όχι. Περνάμε στις ψηφοφορίες λοιπόν. Άρθρο 1. Συμβασμός Α. Τεσσάρων πολιτικών ομάδων. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 2. Παράγραφος 1. Συμβασμός Β. Δύο πολιτικών ομάδων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 2, παράγραφος 3, 2 ε, του εισηγητή υπέρ, κατά αποχές ε, νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 2, αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία, ωραία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Έντεκα υπέρ, 23 κατά. Άρα απορρίπτεται, καταφανώς. Δύο του εισηγητή υπέρ, μα μόλις την ψηφίσαμε κυρία Μπερές. Μόλις την ψηφίσαμε.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 2. Τσαμπαωρή. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 11. Χάιντ Μπέκερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 3, παράγραφος 1, μία προφορική έχουμε εδώ, τροπολογία, ε, αντί για equally, equal partnership, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά αποχές θα επαληθεύσουμε την 13, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, 17 υπέρ, κατά 14, τέσσερις αποχές, απορρίπτεται. Εγκρίνεται, διορθώνει η πρόεδρος. Άρθρο 4, παράγραφος 1, τροπολογία 4, Τσάμπα ουρί με μία προφορική, δεν υπάρχει αντίθεση στην προφορική, ψηφίζουμε ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 5, τροπολογία 14 της κυρία Βαλτακίνο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε. Επαληθεύουμε την 5. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 17 υπέρ, κατά 16, καμία αποχή, εγκρίνεται. Τροπολογία 6 της κυρίας Μπαλτακίνο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 της ιδίας υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται ψηφίσουμε το σύνολο του, της ενδιάμεσης έκθεσης ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 32 υπέρ, κατά 3, ε, καμία αποχή. Εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε την έναρξη διαπραγματεύσεων Ποιο επιθυμεί τι διαπραγματεύσει παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν είναι έτοιμο και εγώ θα ήθελα να ζητήσουμε εντολή στην Ολομέλη επί του θέματος αυτού γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να βελτιστοποιήσουμε το πλαίσιο οργάνωσης αυτής της εντολής. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 21 υπέρ κατά 15. Μία αποχή. Άρα απορρίφθηκε η πρότασή μου. Ε, χρειαζόταν πλειοψηφία 26 ε, συνεπώς ε, θα μπορέσουμε να ζητήσουμε από την Ολομέλεια εντολή για το θέμα αυτό. Euh, Θα ψηφίσουμε τώρα το σημείο 23 πρόκειται για την ε, πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού 718 σε σχέση με την ε, μεταφορική ικανότητα των κοινοτικών στόλων σε εσωτερική ναυσιπλοεία για την ε, πρόθεση των μεταφορών Δια της ε, πλωτής οδού, δηλαδή το περίφημο καμποτάζ. Στο άρθρο 1, στην εισαγωγή του αρχικού κειμένου υπάρχει η τροπολογία 3 της ηγήτριας υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 19 υπέρ, κατά 18, καμία αποχή. Εγκρίνεται με μία ψήφο. 11 Σρέτερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Στο άρθρο 1, στην Παύλα 2, συμβασμός α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Β στο 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Στο 4-7 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά αποχές θα υπαλληθεύσουμε ηλεκτρονικά, αλλά νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Ψηφίσατε όλοι. Δεκαεπτά υπέρ, δεκαοκτώ κατά, μία αποχή. Απορρίπτεται λοιπόν. Ως προς τις απαλλαγές Λυπάμαι, λυπάμαι, κάνω συνεχώς λάθη σήμερα. Στο 4, τροπολογία 14, καταπίπτει. Όχι, όχι, δεν τα καταφέρνω σήμερα. Ξαναρχίζω. Η 7 απορρίφθηκε, άρα θα ψηφίσουμε την 14, Φιλίπ Ντεμπάκερ, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Στο 5 τροπολογία 8 της εισηγήτριας υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 15 μπορούμε να ψηφίσουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 είναι μη αποδεκτή στο 2-9 της κυρίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το, την, την αιτιολογική σκέψη 6, τροπολογία 1, τη, μία, της εισηγήτρες, με συγχωρείτε. Ψηφίζουμε την ε, πρώτη τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 8 λέει η πρόεδρος καταπίπτει. Άρα ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 34 υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή. Άρα η γνωμοδότηση της κυρίας Γιούτα Στάινρουκ εγκρίθηκε. Φτάνουμε τώρα στις απαλλαγές και ψηφίζουμε καταρχήν την απαλλαγή για το τμήμα 3 της Επιτροπής για τον γενικό προϋπολογισμό. Στην παράγραφο 1 έχουμε τροπολογία 1 του Τσαμπαωρή, η συγκήτρια είναι υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στην παράγραφο 6 έχουμε το συμβασμό α τεσσάρων πολιτικών ομάδων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οι 2 και 3 καταπίπτουν, άρα ψηφίζουμε το σύνολο της, ε, του κειμένου ηλεκτρονικά, αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 34 υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή, άρα εγκρίνεται. Τώρα... Περνάμε στο σημείο 25, απαλλαγή Πρώτα στα 29. για τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών. Ένα, υπέρ κατά, ε, εγκρίνεται. Τρία, συμβαστική τέσσερα, από τέσσερις ε, πολιτικές ομάδες, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικά, έναρξη. Όλοι ψήφισαν πέρας. 33 υπέρ, 3 κατά, 0 αποχές. Εγκρίνονται λοιπόν η απαλλαγή. Σημείο 25. Απαλλαγή σε ό,τι αφορά τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς για την ε, κατάρτιση. Παραγράφη 2 της Επιλογίας 1 της Χάρκιν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Τροπολογία 2 της κυρίας Χάρκιν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5. Ε, Έχουμε προφορική ε, τροπολογία. Adopting a formal decision, the governing board failed to inform the parliament of its, of its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 provided in the regulation. Δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Ας ψηφίσουμε λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση για να στείλουμε ένα καλό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έναρξη. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. 37 υπέρ ηλεκτρόεδρος, 30... 35 υπέρ, μία ψήφος κατά, 0 αποχές. Επομένω ελπίζω να ακούσει η Επιτροπή το μήνυμα ε, της ε, Επιτροπής μας, ε, επί το συνόλου της νομοδότησης τώρα, υπέρ, ή μάλλον έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας, 32 υπέρ, 3 κατά, 0 αποχές. Περνάμε στο σημείο 26, απαλλαγή 2012 του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθήκων Διαβιώσεων και Εργασίας. Για το σύνολο της απαλλαγής ηλεκτρονικά έναρξη. Πέρας. 33 υπέρ, 3 κατά 0 αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στο σημείο 27, απαλλαγή για το... Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνδικών Διαβιώσεων και Εργασία. Στην παράγραφο 1 πρέπει να ψηφίσουμε τέσσερι ε, τροπολογίε ε, από κοινού. Ουσιαστικά πρόκειται για μία τροπολογία που αφορά τέσσερις παραγράφους. που έχει ως στόχο την εναρμόνιση των ε, ευρωπαϊκών προσόντων. 1, 3, 4, 7 που αφορούν τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4. Τέσσερις ε, τροπολογίες του Σεργίου κουτιερε Πριέτο. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 1. Τροπολογία 1 της κυρίας Χάρκιν. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Τροπολογία 5 της ίδιας. Ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Τροπολογία 6 του όρη. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 5. Τροπολογία 8 του Σέργιο Κουτιέρε Βιέτο. Υπέρ κατά Αποχές. Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Για το 8. Πέρας. 21 ψηφί υπέρ, 15 κατά, 0 αποχές. Εγκρίνεται. Επί του συνόλου της νομοδότησης ηλεκτρονικά. Έναρξη. Πέρας. 33 υπέρ, 3 κατά, 0 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. Περνάμε στο τελευταίο σημείο που αφορά απαλλαγή, σημείο 28, 2012, για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΕΝΤΕΦΟΠ. Παράγραφος 1, ε, τροπολογία 1 της Χάρκιν. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3, ε, τροπολογία 2, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5, συμβαστική α από 4 πολιτικές ομάδες. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επί του συνόλου ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Υπέρ, ναι, συγγνώμη, έναρξη. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ναι. Τα αποτελέσματα. Θα σας ενδιαφέρουν λογικά. 31 υπέρ, 4 κατά, 0 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. Περνάμε στο σχέδιο γνωμοδότησης που η Επιτροπή μας ε, εκπώνησε για την Επιτροπή Προπολογισμού για τις υπερματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Διδάγματα που πρέπει να αντιληφθούν και μελλοντικέ προοπτικές. Παράγραφος 1. Τροπολογία 1 του Τζιν Λάμπερτ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 2. Ε, Συμβαστική ε, τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6. G. Lambert. Υπέρ κατά αποχές Ας επαληθεύσουμε για την τροπολογία 6. Έναρξη. Πέρα. 19 υπέρ, 14 κατά, 0 αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφο 4. 7 τη υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφο ε, τροπολογία μάλλον, 8 Λάμπερτ υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφο 5. Τροπολογία 9 Λάμπερτ υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 10 της ηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 Χάρκιν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5. Τροπολογία 12 Λάμπερτ και Μπεναραπατού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 συμβαστική Β από τρεις πολιτικές ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινού το σύνολο των τροπολογιών 16 έως 30. Όχι. Πού θέλετε να σταματήσουμε. Εντάξει. Δεν θα λέω όμως τις παραγράφους, μόνο τις ε, τροπολογίες, όλες είναι τις συζυγήτριες. 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20. Α, ας επαληθεύσουμε τη 19. Ηλεκτρονικά. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αφού ξέρω ότι έχει εγκριθεί, θα δείτε. 19 υπέρ, 13 κατά μηδέν αποχές. Συνήθως ο αντιπρόεδρος ε, παρακολουθεί πολύ καλά. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές Θέλετε να παληθέψουμε κύριε Μάν. Παρακαλώ. Για την 22.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 Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. «29 υπέρ, 4 κατά, 1 αποχή». Ε, με εκπλήσει βέβαια η τροπολογία που απορρίψατε που αφορά την διαπραγματευτική ικανότητα του Κοινοβουλίου. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για το σημείο 20. Ψηφίζουμε την έκθεση πρωτε... πρωτοβουλίας για μια μελέτη για τις ε, δραστηριότητες και το ρόλο της ΕΤΡΟΙΚΑ, δηλαδή της Επιτροπής του Διεθνούς Ομοσπονδιακού Ταμείου και της Κεντρικής Τράπεζας, ε, για τις ε, χώρες που μπήκαν σε πρόγραμμα διάσωσης στην Ευρωζώνη. Πρόκειται για μια έκθεση για την οποία συγητής είναι ο κύριος Σέρκας και συνάδελφος Βεστρέγια νομίζω ότι έχει ένα ζήτημα επί τη διαδικασία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω να αποσυρθούν οι δικές, μας οι δικές μου τροπολογίες 106, 116, 170, 185, 241, και 243. Ευχαριστώ πολύ. Να αποσυρθούν αυτές οι έξι τροπολογίες, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Είναι Πάστος. Και εγώ θα ήθελα να αποσύρω τις τροπολογίες μου 109, 129 και 181. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θέλει να αποσύρει τροπολογία. Όχι. Όλα τα υπόλοιπα θα τα ψηφίσουμε λοιπόν. Παράγραφος 1. Συμβαστική δέλτα από 4 σώματες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Συμβαστική F ε. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 45. Αποσύρθη. Στην πράγραφο 3 έχουμε τη συμβαστική Z από δύο ομάδες. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Μετά. Συμβαστική Α4. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική G. Υπέρ, κατά, αποχές ηλεκτρονικά για το G. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 25 υπέρ, 8 κατά 0 αποχές. Πολύ ξεκάθαρο αποτέλεσμα, εγκρίνεται. Η 50 απεσύρθη. Μετά 51 καλύπτεται. Περνάμε λοιπόν στην παράγραφο 4, συμβαστική H, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική I. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 69 επεσήρθη. Πάμε λοιπόν στην 70. Τζούμπερ και Μέρφυ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική Κάπα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 72 καταπίπτει. Περνάμε λοιπόν στη συμβαστική σήμα S. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική J. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική λάμδα L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 Μέρφυ και Ζούμπερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική FF υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Υπάρχει πρόβλημα. Κύριε Σιγητά. Εκτός μικροφώνου. Tout va bien. Alors, merci de votre vigilance. Άρα, ευχαριστώ. Ε, 90. Τσούπερ και Μέφη. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική ταφ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική εμ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Η 95 καταπίπτει. Πάμε στην 7 λοιπόν. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 106 εστρέλια. Απεσύρθη. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα για την παράγραφο 8. Συμβαστική π. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πολλές εδώ καταπίπτουν και περνάμε στην 112. Μέρφυ και Τζούμπερ. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 116 απεσύρθη. Πάμε στην συμβαστική U. Υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Σεβαστική Q. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εκατόν συγγητρίας υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά, 128 127. Μέρφυ και Ζούμπερ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 128. Το κύριο Πουπάκη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 129. Απεσύρθη. 131. Της κυρίας Ράπτη υπέρ. Κατά. Αποχές. Να δούμε ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονική επαλήθευση έναρξη. Πέρας. 21 υπέρ, 15 κατά. 0 αποχές. Εγκρίνεται. 132 της κυρίας Κορνελίσεν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 133 του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 142, Ζούμπερ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 145 Μέρφυ και Τζούβερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 146 των ιδίων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 147 Πολ Μέρφυ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 148 Κοστέλο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 13. 149 καταπίπτει. Μπλα μπλα μπλα λέει πρόεδρος. 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 153 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβιβαστική Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 155 το ΕΛΚ εδώ θέλει ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα μέχρι το Health for Everyone, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Εντάξει, ας επαληθεύσουμε για το πρώτο τμήμα. Πέρας. 20 υπέρ, 16 κατά, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα Περ. Κατά. Αποχές. Το δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. 156 χάρκεν. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 157 ζητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 158 καταπίπτει. 159. Εστρέλα. Δεν απεσύρθη. Σε δύο τμήματα λοιπόν. Υπέρ του πρώτου τμήματος, χωρίς την υποσημείωση. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Για την υποσημείωση. Υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική W. Υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 164. Τζούμπερ Μέρφυ. Υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 163 βάστος υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 165 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 167 Μέρφυ Ζούμπερ υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 170 επεσήρθη. 176 του εισηγητή με προφορική τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την 176, όχι. Ας ψηφίσουμε λοιπόν 176 υπέρ κατά αποχές. Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε πέρας. 17 υπέρ, 18 κατά, 2 αποχές. Δεν εγκρίνεται λοιπόν, απορρίπτεται. 177 τζούμπερ υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 178 μέρφυ υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 181 βάστος υπέρ. Α, απεσύρθη. Συγγνώμη. 182 παραμένει υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 183 καταπίπτει, 184 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 185 μάλλον απεσύρθη τα έξι κατατμήματα. Ψηφορία κατατμήματα λοιπόν. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και το υπόλοιπο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Α, σε το δεύτερο τμήμα. Έναρξη. Πέρας. 17 υπέρ, 19 κατά, 0 απόχέ. Είχατε δίκιο, απερίφθη. 19 συμβαστική αλφα υπέρ, κατά απόχέ εγκρίνεται. Πρέπει να ψηφίσουμε τα 187 πρώτα. Υπέρ, κατά απόχέ απορρίπτεται. 193 Τζούπερ, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική εισήγηση. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρεις τροπολογίες ε, της Τζούπερ. Να τις εξετάσουμε με από κοινού. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική BB, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. ...204 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 214 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Ας Πέρας. 30 υπέρ, 7 κατά. Δεν είχα δει αυτό πάντως εγώ. 215 καταπίπτει. απερίφθη, ή μάλλον επεσήρθη η τροπολογία Μπενιών. Πάμε λοιπόν στη βασική DD, υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Μόνο μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε την DD, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική ε, ε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Διακόσια 27 μάλλον. Υπέρ κατά απορρίπτεται. 228 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 233. Πολ Μέρφυ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 235 Κονέλισεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 235. Πέρας. 29 υπέρ, 4 κατά, 2 αποχές. Συμβαστική GG. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 2.37 το σύγητη υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 2.39 καλύπτεται από τη συμβαστική. 2.40 υπέρ κατά, αποχές, απορρίτεται. 2.41 στρέλα υπέρ, απεσύρθη. 2.42 το σύγγεται υπέρ, κατά, αποχές, εγκρινέται. 2.43 επίσης απεσύρθη. 2.44 υπέρ, κατά, αποχές, υπέρ της 2.44. Κατά. Απορρίπτεται. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αν έρθετε στη θέση μου θα δείτε τέλος πάντων. Ας επαληθεύσουμε. εντάξει δεν είμαι και στα καλύτερα μου σήμερα, αλλά ούτε και κάποιο από εσάς είναι. Λοιπόν, ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 29 υπέρ, 7 κατά, 0 αποχές. Μεγάλη επιτυχία της τροπολογίας έλυσαν. Περνάμε λοιπόν στα σημεία 1 33. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την ατολική σκέψη α στη 10. Α, συγγνώμη. Μετά το 1β Μετά το 1 έχουμε την τροπολογία 1 της Κονέλισεν. Υπέρ κατάποχες Και πάλι μεγάλη επιτυχία η κυρία Κορνέλησεν. Περνάμε λοιπόν στην 10 Τσούμπερ. Τρία του εισηγητή. Μετά τα υπόψη 1. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Τέσσερα του εισηγητή. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Να σας πω κάτι. Οι 7 έως 9 καταπίπτουν. Συμφωνείτε όλοι. Ωραία, εξαιρετικά. Μετά όμως πρέπει να ψηφίσουμε το 10. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Μετά από το υπόψη α, 11, 12 και 13 καταπίπτουν. Συμφωνούμε. Τέλεια. 14. Τσούπερ υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Συμφωνούμε. Ωραία. 15. Φωτανία υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Συμβαστή Β. Κοστέλιο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 17 Κοστέλιο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά αποχές υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β. Υπέρ. Ας επαληθεύσουμε. Για τη 19. Γιατί δεν είμαι σίγουρη για τίποτα σήμερα. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία, πέρας. 21 υπέρ. 14 κατά. 0 αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Β. Υπέρ κατά αποχές γκρίνεται. Συμβαστική σε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27 βενιό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ας ψηφίσουμε τώρα επί του συνόλου της έκθεσης για τον ρόλο και τις δραστηριότητε της Τρόικα. Υπέρ, συγγνώμη, έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ψηφίσατε όλοι, πέρας. 27 υπέρ, 7 κατά, 2 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ωραία. Τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Ησυχία παρακαλώ. On va suspendre notre séance une minute. Διακοπή ενός λεπτού. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας, διότι μόλις ήρθε η συγγήτρια. Έχω ένα κακό νέο βέβαια, γιατί θα πρέπει να διακόψουμε μετά, γιατί είχαμε ε, προβλέψει μία σύνοδο ψηφοφοριών πολύ μακρύτερη και για όλα αυτά φταίει ο Αλεχάνδρο Θέρκας ο οποίος είναι πολύ καλός ε, διαπραγματευτής. Άρα θα ψηφίσουμε, ε, αντί να ψηφίσουμε 244 τροπολογίες, ψηφίσαμε τροπολογίες συμβιβασμού που προχώρησαν ε, με γοργούς ρυθμούς. Γι' αυτό μετά το 16 θα διακόψουμε και θα περιμένουμε τους προσκαλεσμένους μας. και θα σας πω δύο λόγια για αυτούς πριν. Λοιπόν, στο 16 πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο δεν μας απασχόλησε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά είναι ύψη της ε, σημασίας, διατεφορά τους όρους εισόδου και διαμονής υπηκών τρίτων χωρών στο πλαίσιο των ε, ενδοεπιχειρησιακών μεταθέσεων. Συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών και στις 5 Δεκεμβρίου του 2011 είχαμε αναθέσει εντολή στους διαπραγματευτές μας. Είναι παλαιά υπόθεση λοιπόν. Τα πράγματα όμως κινούνται αρκετά το, θέμα αυτό ήταν εν περιμέναμε τη, θέση του Συμβουλίου για την οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους, γι' αυτό και περιμέναμε τόσο πολύ. Αλλά τα πράγματα κινούνται εκ νέου και θα δώσω το λόγο στη Λίζα Γιάκονσάρη για να μας πει πού βρισκόμαστε και πώς, ε, τι διεμήφθη μάλλον στον χτεσινό τριμερή διάλογο. Η Σάρι είναι από το ΕΛ και η κυρία Χίρς από εμάς, Ελίζαβετ Σρούτερ από τους ε, Πράσινους, Τόμας Χάντελ από την ΚΟΕ, ECR, Ρότζερ Έλμερ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όπως είπατε, χθες πραγματοποιήθηκε ένας ε, τελικός τριμερής διάλογος ε, για την οδηγία για τις ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις. Ε, τις τελευταίες εβδομάδες προσπαθήσαμε μαζί με τους κοιόδες συζητητές να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό με το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο δεν συνεργάστηκε ιδιαίτερα επικοδομητικά. Η Κομισιόν ήταν πιο διατεθειμένη να βρει ένα συμβιβασμό. Όπως γνωρίζετε, η αρχική μας θέση ήταν η ίση μεταχείριση και να διαγράψουμε την αναφορά του, της Κομισιόν και του Συμβουλίου στην ε, πολύ επίμαχη νομοθεσία για την απόσπαση των εργαζομένων. Ήταν πολύ ισχυρή αυτή η εντολή μας οι περισσότερες ε, πολιτικές ομάδες ε, την υποστήριξαν ε, στην Επιτροπή μας. Αυτό εξηγεί ακριβώς ότι το να, αυτό, το να δεχτούμε αυτό που απορρίψαμε νωρίτερα δείχνει πόσο ανοιχτοί είμαστε. Ωστόσο, ζητήσαμε από το Συμβούλιο να επανέλθει στην αρχική πρόταση που επιβεβαίωνε τουλάχιστον την ίση μεταχείριση όσον αφορά την αμοιβή. Το άρθρο 18 που έχει να κάνει με τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις ε, συνθήκες εργασίας ε, συμπεριλαμβανομένων ε, των συνθήκων που έχουν να κάνουν με την υγεία και την ασφάλεια. Το Συμβούλιο δέχτηκε μόνο την ίση μεταχείριση όσον αφορά την αμοιβή. Στο άρθρο 5 που σχετίζεται με τα κριτήρια εισδοχής ο εργαζόμενος δεν μπορεί να προσφύγει σε δικαστήριο για τα δικαιώματά του ε, ε, μόνο με τις ε, διοικητικές διαδικασίες των κρατών μελών και όχι να θεωρούνται δεδομένα τα ίσα, δεδο... ε, ίσα τα δικαιώματά του. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι πρόκειται για εξειδικευμένους εργάτες. Δεν μιλάμε για ανειδίκευτούς όταν μιλάμε για ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις. Τα κριτήρια εισδοχή ε, δεν προβλέπουν προσφυγή σε δικαστήριο. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Το Συμβούλιο ε, επίσης προτείνει η αναδιατύπωση του εκτιμώντα 11, τη αιτιολογική σκέψη 11. Αλλά αυτό μάλλον είναι κοσμητικό θέμα. Νομίζω ότι η λύση αυτή επιφέρει περισσότερη σύγχυση όσον αφορά τα δικαιώματα των ε, εργαζομένων ε, που ε, κάνουν ενδοεπιχειρησιακή μετάθεση. Δεν είναι καλός ο συμβιβασμός αυτός και το Συμβούλιο δεν καταβάλει καμία προσπάθεια να βρεθεί ένας καλύτερος συμβιβασμός. Ζητώ λοιπόν από την Επιτροπή να μου πει ως εισηγήτρια τι μήνυμα να στείλω προς την Προεδρία. Ως Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσουμε εάν αυτή είναι μια καλή βάση για να κλείσουμε τις διαπραγματεύσεις ή χρειαζόμαστε ότι θα πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες στο Συμβούλιο. Ο χρόνος είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος να αναβληθεί το όλο θέμα για μετά τις εκλογές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό δεδομένου ότι η Προεδρία δεδομένου ότι αυτή η συμφωνία έχει προς το παρόν την έγκριση του Συμβουλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους για τη σκληρή δουλειά που έχουν κάνει τις τελευταίες εβδομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Άρα ε, φαίνεται ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τους εποχικούς. Είχαμε επιτυχία, το ίδιο αφορά ε, τους αποσπασμένους, αλλά εδώ δεν πάνε και τόσο καλά τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι οφείλεται στην ομάδα διαπραγμάτευσης ε, του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου. Σάρι Εσάγια και μετά ποιος άλλος θέλει το λόγο. Ησυχία. Ακολουθώ τον κατάλογο. Σάρι Εσάγια, κυρία Χίρς, η Ελίζαμπετ ε, Σρετέρ, Αλεχάνδρο Θέρκας. Αυτά προς το παρόν. Σάρι Εσάγια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με την εισηγήτρια Λίσα κονσάρι. Ήταν δύσκολε οι διαπραγματεύσει αυτές, οι διαπραγματεύσει των τελευταίων εβδομάδων. Και πολύ δύσκολο είναι το γεγονός ότι έχουμε μόνο μοιρασμένε αρμοδιότητες σε αυτά τα πολύ κεντρικά ζητήματα, τα οποία είναι τα βασικά αυτού του νομοθετήματος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Λίζα για την σκληρή δουλειά της και να ευχαριστήσω και τους άλλους σκιώδεις εισηγητές. Προσπαθήσαμε να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν όταν μεταφέρθηκε το θέμα της αμοιβή στο άρθρο 5, διότι το άρθρο 5 δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. παρότι είναι ένα θέμα που συνδέεται στενά με τα θέματα της δικής μας Επιτροπής. Από τεχνικής άποψης λοιπόν ε, μας δυσκολεύει αυτό, διότι το Συμβούλιο δεν μετακινείται καθόλου όσον αφορά τις θέσεις του. Και έτσι έχουμε φτάσει στο σημείο που θα πρέπει να εξετάσουμε αν είναι πιο σημαντικό να ολοκληρώσουμε τις εργασίες τώρα με μεγάλη πίεση χρόνου ή θα προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση, έναν καλύτερο συμβιβασμό δηλαδή. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων Περίεργο ήταν ότι από την Προεδρία λαμβάναμε προτάσεις οι οποίες κατόπιν αποσύρονταν. Είχαμε δηλαδή οπισθοχώρηση του Συμβουλίου από τη θέση που μας ε, είχε παρουσιάσει επανειλημμένα και αυτό μας μπέρδεψε χθε. Λάβαμε τη νέα διατύπωση του άρθρου 5 και σήμερα το πρωί λάβαμε μία δήλωση της Επιτροπής. η πολιτική μου ομάδα αναρωτιέται τι θα πρέπει να κάνουμε στην περίπτωση αυτή, αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε να συνεχίσουμε με τις διαπραγματεύσεις, διότι δεν υπάρχει μόνο αυτό το θέμα, έχουμε και άλλα δύο, τις διμερείς ε, συμφωνίες και θέματα κοινωνικής ασφάλισης που εκκρεμούν όσον αφορά τη δική μας Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω λέγοντας ότι πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ολοκληρωθούν οι εργασίες αυτές. Δεν ξέρω όμως ποιο θα είναι το τίμημα που θα πρέπει να πληρώσει η Επιτροπή μας. Αλλά ε, εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να φτάσουμε να το απορρίψουμε. Όπως είπε η Λίσα όμως δεν είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τη διατύπωση και ιδιαίτερα όχι με την αιτιολογική σκέψη 11. Δεν μας προσθέτει τίποτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Ήταν δύσκολες οι διαπραγματεύσεις. Χαίρομαι και εγώ όμως που χθες το ΕΛΚ δέχτηκε να συνεργαστεί, διότι κατά τη γνώμη μας είναι πολύ σημαντικό να πετύχουμε συμφωνία με το Συμβούλιο στο θέμα αυτό. Αυτό είναι το ερώτημα που θα πρέπει να θέσουμε. Δεν είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι. Πιστεύω όμως ότι θα ήταν λάθος ε, μήνυμα το να μην ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις. Διαπραγματευόμαστε εδώ και 1,5 χρόνο, δύο χρόνια το οποίο σημαίνει ότι δεν πρόκειται να βελτιωθεί η κατάσταση. Υπάρχουν διαφορετικές θέσεις, διστάμενες θέσεις και τελικά το να πούμε ότι θέλουμε να στείλουμε ένα σαφές ευρωπαϊκό μήνυμα προς τα τρίτα κράτη όσον αφορά τις ε, ε, ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις. Ε, νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό παρότι μπορεί να υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία να μην είναι ιδανικά κατά τη γνώμη μας. Το ζήτημα είναι λοιπόν Δεν πιστεύω ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση, πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο ώστε να ολοκληρώσουμε το θέμα και να δείξουμε ότι ως Ευρωπαίοι ε, βρίσκουμε πάρα πολύ σημαντικό αυτό το σύμπλεγμα θεμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ η Ελίζα Πεθσέντερ. Και η δική μας ε, πολιτική ομάδα ε, εξετάζει τα τελευταία αποτελέσματα. Η Τζιν είναι και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ εξετάζει το θέμα αυτό. Εμείς το βλέπουμε από την πλευρά της Επιτροπής Απασχόλησης. Στο κάτω-κάτω θα πρέπει να κοιτάξουμε γιατί έχουμε το νομοθέτημα αυτό. Πρόκειται για βελτίωση. Επί της ουσίας υπάρχουν κάποιες ε, ομάδες ανθρώπων που Αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες όταν περνάνε από τη μία χώρα τη ευρωπαϊκή Ένωση στην άλλη και θέλουμε να μειώσουμε αυτό το άχθο. Δεν θέλουμε όμως ε, να ε, του δώσουμε ε, λιγότερα δικαιώματα και αυτό ακριβώς έχει συμβεί. θα είχαν αυτοί οι άνθρωποι πολύ καλύτερα δικαιώματα εάν δεν είχαμε την οδηγία αυτή. Ουσιαστικά δηλαδή πιέζει προς τα κάτω τα δικαιώματά του και για μένα αυτό είναι το αποτέλεσμα. Στην τελευταία πρόταση έχουμε μια μικρή βελτίωση, αλλά το τελικό αποτέλεσμα ε, είναι μάλλον μείωση. Θα έχουν μόνο τα δικαιώματα μετατιθέμενων εργαζομένων, ε, τα οποία είναι πολύ λιγότερα από ό,τι έχουν αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχουν ε, τα δικαιώματα των εργαζομένων και αυτή η οδηγία έχει να κάνει με την κινητικότητα, όχι με την ελευθερία παροχή υπηρεσιών. Ε, ρυθμίζουμε λοιπόν εδώ θέματα ε, ε, ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται καθόλου από τη συνθήκη. Αλλά τώρα σε αυτή την πλεγμένη δομή συμπεριλαμβάνουμε άλλη μία ομάδα που κατά τα άλλα υπόκειται στην ελεύθερη κινητικότητα. Και έτσι είχαμε αιτιολογήσει αυτή την οδηγία και τώρα τα μπερδεύουμε όλα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολη, πολύ μπερδεμένη αυτή η δομή που περισσότερα προβλήματα μας δίνει από ό,τι πλεονεκτήματα και για τους ανθρώπους που αφορά αυτή η οδηγία τελείως νυφάλια θα πρέπει να σκεφτούμε γιατί υπερψηφίζουμε μία οδηγία που ε, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε καλύτερη θέση τους ε, επιδεινώνει τη θέση τους. Τι κέρδος έχουν από αυτήν. Εάν δηλαδή δεν έχουμε το νομοθέτημα αυτό, είναι σαφή τα δικαιώματά τους, έχουν τα δικαιώματα που απορρέουν από την ελεύθερη κινητικότητα, έχουν δηλαδή ε, ίσα δικαιώματα με τους άλλους εργαζομένους. Γι' αυτό εμεί βλέπουμε επικριτικά το θέμα αυτό. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα τη θέση μα. δεν έχουμε οριστικοποιήσει ακόμα τη θέση μας, ε, αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει προστιθέμενη αξία ούτε με την τελευταία πρόταση του Συμβουλίου. Κατόπιν έχουμε αυτή την δήλωση που έχει να κάνει με τι διμερείς συμφωνίε. Υπάρχουν τέτοιε. Ανάμεσα στην Ισπανία και το Μεξικό, για παράδειγμα. Υπάρχουν εδώ διμερεί ζητήματα, ε, υπάρχουν διμερεί συμφωνίε όπου ρυθμίζονται κάποια ζητήματα. Θα πρέπει με βάση αυτή την οδηγία να εξεταστούν αυτέ οι συμφωνίε. Δηλαδή, πολύ καλύτεροι κανόνε θα επαναξεταστούν με βάση αυτή την οδηγία, μήπω τυχόν και είναι υπερβολικά καλέ οι, οι, οι ρυθμίσει αυτέ. Έτσι καταλαβαίνω εγώ τον έγγραφο τη Κομισιόν. Και αυτό το βρίσκω οξύμορο. Εάν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες και αναφέρεται εδώ η ε, επιστροφή ε, συντάξεων στο Μεξικό ή ε, κοινωνική ασφάλιση στο Μεξικό. Αυτά είναι τα αντικείμενα αυτής της διμερούς συμφωνίας. Με την οδηγία αυτή τα μπλέκουμε όλα και επίσης μειώνουμε τα δικαιώματα. Αυτή η δήλωση για μας δεν αρκεί. διότι ακριβώς ε, τις ε, σημαντικές περιπτώσεις ε, τις δυσκολεύει πάρα πολύ και αμφισβητούνται οι καλές διμερείς συμφωνίες. Η πολιτική μας ομάδα θα συνεχίσει να το συζητάει αυτό τις επόμενες ώρες, αλλά αμφιβάλλω αν θα υπερψηφίσουμε το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ο Αλεχάνδρο Φέρκας, καταρχήν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εντάχει, και με σαφήνεια θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελίσσα διότι ήταν ιδιαίτερα ευέλικτη. Αλλά θα ήθελα να πω ότι δεν έχω δει άλλη τέτοια διαπραγμάτευση, δηλαδή το Συμβούλιο ε, απέριψε όλες μας τις ε, προτάσεις και παλινοδεί σε σχέση με την αρχική του προσφορά. Άρα δεν είναι αυτή η είναι επιβολή θέσεων και πολιτικά είναι απαράδεκτο και ακόμα και νομικά δεν θα επιλύσει κανένα ζήτημα. Δεν μπορούμε να αποσύρουμε το άρθρο 14 και να βασιστούμε στο άρθρο 5 πού βρίσκονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να κάνουν ό,τι θέλουν, διότι όταν ισχύσει το άρθρο 5, τότε οι γιούροι η Λίμπε θα πρέπει να διαπραγματευτεί και θα είναι και η μόνη που θα μπορεί. Αλλά αυτό είναι πολύ μακριά από την αρχική μας ε, πρόταση σε σχέση με τους αποσπασμένους και την ε, ισότητα μεταχείρισης γιατί το Συμβούλιο δεν μας δίνει τίποτα. Νομίζω ότι η θέση της σοσιαλιστικής ομάδας είναι να πούμε ότι δεν δεχόμαστε μία τέτοια στιγνή επιβολή κατά της πολιτικής, κατά της ε, ε, νομικής ε, λογικής. Μα δεν μπορούμε να έχουμε μία οδηγία η οποία να είναι ένα κενό γράμμα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει ε, να μην υπάρχει σπουδή. Δηλαδή, την τελευταία στιγμή μας διαβουλεύονται διαφορετικά, δεν θα υπάρχει ε, οδηγία. Εμείς θα δεχτούμε μόνο ως βάση το άρθρο 14 και δεν μπορούν να μας επιβάλλουν κάτι την τελευταία στιγμή. Δηλαδή, δεν θα μπορέσουμε να δεχτούμε μια τέτοια συμφωνία και θα ε, προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αν χρειαστεί. Thank you, Madam President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν με προβληματίζουν καθόλου οι λεπτομέρειες αυτού του ζητήματος ε, για την απόσπαση εργαζομένων. Αυτό που με προβληματίζει είναι η ε, υποβόσκουσα τάση που υπάρχει. Οι υπήκοοι των τρίτων χωρών δεν θα έχουν πλήρη δικαιώματα όταν θα πηγαίνουν οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό δείχνει και την ίδια τάση που, ε, που σε ένα κείμενο που είχαμε λάβει πέρσι τον Απρίλιο. Τότε λέγαμε λοιπόν ότι όταν οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι πήκοοι ε, πάνε να δουλέψουν σε άλλη χώρα, τότε θα πρέπει να πάνε σε εκείνους και όχι σε οποιονδήποτε άλλο φορέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν είναι εχθρική τάση δική μου απέναντι σε αυτούς τους υπηκόους. Πρέπει να μάθουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Γιατί, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους, με τις υπόλοιπες ε, χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς έχουμε αυτή την κοινοπολιτεία που συμπεριλαμβάνει το 1 τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού. Ε, παλιότερα ήταν αυτοκρατορία. Βεβαίως ε, έχουν περάσει αυτές οι ημέρες ε, και δεν λέω ότι είναι καλό ή κακό το να έχουμε αυτοκρατορία. Όμως όλες αυτές οι χώρες χωρίς καμία εξαίρεση εθελοντικά προσχώρησαν στην Βρετανική Κοινοπολιτεία με επικεφαλής τη Βασίλισσα. Από εκεί πέρα λοιπόν οφείλουμε και έχουμε υποχρέωση ε, να τους σεβαστούμε και να τους τιμήσουμε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο. Και πάλι βλέπουμε ότι θα τύχουν αρνητικής διάκρισης. Είμαστε μικρή χώρα, βεβαίως η πολυπληθέστερη σε πυκνότητα πληθυσμού στην Ευρώπη και παρόλα αυτά με τέτοιους κανονισμούς αναγκαζόμαστε να δεχόμαστε υπηκόους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θεωρώ ότι ε, έχουμε χρέος τιμής ε, και ευγνωμοσύνης προς τους υπηκόους αυτών των τρίτων χωρών που είχαμε κατακτήσει στο παρελθόν. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε υπό ευρωπαϊκούς ε, κανονισμούς να κάνουμε αρνητικές διακρίσεις εναντίον των επικών της κοινοπολιτείας, γιατί αυτό, περί αυτού πρόκειται, αυτή την παρατήρηση έκανα πέρυσι τον Απρίλιο, κανένας δεν απάντησε στην παρατήρησή μου ότι πρόκειται για αρνητική διάκριση που απαγορεύεται βάσει της ηθικής Λισαβόνας και θέλω να μου πείτε γιατί επιτρέπεται αυτή η διάκριση. Ευχαριστώ. Θα δώσουμε και πάλι το λόγο στην εισηγήτρια. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιο άλλο τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ κατάλαβα το μήνυμα της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου ότι πρέπει να ξαναξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις και να μείνουμε στενά στην εντολή της Επιτροπής μας και να διασφαλίσουμε την ισότιμη μεταχείριση. Είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και πάλι όμως ε, θεωρώ ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό γιατί είναι πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο να μην ε, αναβάλει αυτή την πολύ σημαντική οδηγία. Προσπαθούμε να πούμε σε επαναδιαπραγμάτευση ιδιαίτερως ε, με το Συμβούλιο και ξεκινάμε απευθείας. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ο κύριος Κλάρκ συμφωνεί απολύτως μαζί σας. Ελπίζω ε, να υπάρχει ίδια στήριξη σε ό,τι φορά την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. Όμως ε, σε αυτό τον φάκελο θεωρώ ότι στο, το σύνολο των πολιτικών ομάδων ε, στηρίζει την εισηγήτρια να διατηρήσει δηλαδή την θέση της Επιτροπής Απασχόλησης στις διαπραγματεύσεις που γίνονται με την ε, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και το Συμβούλιο σε αυτή τη φάση. Με την ελπίδα να βρούμε μια καλύτερη συμβιβαστική λύση σε σχέση με αυτή που έχουμε σήμερα επιτάπητος. Ε, εντάξει, θα σταματήσουμε εδώ σε ό,τι αφορά αυτό το σημείο της ημερήσης διάταξης και επενθυμίσω ότι στις 11.30 έχουμε τα απορίσματα μιας πολύ σημαντικής μελέτης ε, που ζητήσαμε από την υπηρεσία μας. Μιας υπηρεσίας που είναι στη διάθεση, ε, στη διάθεσή μας για να αξιολογήσει την προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών θέσεων ε, την οποία Ζητήσαμε λοιπόν για να εξετάσει τα αποτελέσματα του ελάχιστου επιδόματος ανεργίας σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Σας ε, καλώ λοιπόν ε, να έρθετε όλοι εδώ στις 11.30. Η πρόεδρος δεν συγγνώμη από τους ε, διερμηνείς. Λέει ότι δεν είναι ευχάριστο να έχουμε τέτοιες διακοπές. Ο oh, κύριος Στέρικας φταίει βεβαίως.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 Υπότιτλοι AUTHORWAVE τα είναι τελείω. <laughs> Θα το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 Υπότιτλοι AUTHORWAVE Αγαπητοί συνάδελφοι, Α, είναι εδώ η συνάδελφο Ελίζαμπεθ Σρέντερ. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ξέρουμε ότι οι διακοπέ ε, αυτέ των συνεδριάσεων δεν είναι πολύ καλέ. Αλλά μπορούμε πλέον να περάσουμε στο επόμενο ζήτημα που αποτέλεσε αντικείμενο συνεδρίαση ε, τη διάσκεψη των Προέδρων, ε, συγγνώμη, Επιτροπής των Συντονιστών του περασμένου Μαρτίου σχετικά με τα πορίσματα σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή προστεθεμένη αξία για να μπορέσουμε να εκπονήσουμε μια μελέτη για το κόστος της μη Ευρώπης, όπως αναφέρεται, στην απουσία συστήματος ασφάλισης κατά της ανεργίας για τη ζώνη του ευρώ. Θα δώσουμε το λόγο στους τέσσερις εμπειρογνώμονες που θα μας παρουσιάσουν τις δύο μελέτες που εφωνήθηκαν. Να υπενθυμίσω μόνο ότι αυτή η μελέτη προέκυψε κατόπιν πρωτοβουλειών που ε, υιοθετήσαμε για κάποια πολιτικά προγράμματα Βεβαίως βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο που δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει αυτή την πρωτοβουλία, αλλά πραγματοποιήθηκε και αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί έρχεται σε μια πολιτική συγκυρία όπου αυτό το ζήτημα θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων για μια πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση. Θα δώσουμε 15 λεπτό σε κάθε ομιλητή, για κάθε μελέτη. Θα ξεκινήσουμε με την ε, πρώτη ομιλία. Την πρώτη μελέτη που εκπώνησε το ΣΕΦΣ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικών Μελετών. Μύροσλαβ Μπευλαβή και Ηλάρια Μασέλη θα πάρουν το λόγο. Ελπίζω να τα είπα σωστά τα ονόματά σας. Έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την εισαγωγή σας αυτή. Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι πρώτη φορά μιλώ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα, διότι ε, και συμμετέχω στο ΣΕΠΣ, αλλά είμαι και βουλευτής ε, στη Σλοβακία. Ε, ελπίζω λοιπόν να μην σα αποϊδεύσω τώρα που βρίσκομαι στην άλλη μεριά. Ε, να αναφερθώ λοιπόν στο θέμα που θα σας παρουσιάσω σήμερα. Θα παρουσιάσουμε μια απλή προσωμείωση, αυτό που εξετάσαμε, την, ε, το, του κόστους της μη Ευρώπης ε, σε, περίπτωση έλλειψης ενός προγράμματος ασφάλισης ανεργίας. Θα κοιτάξουμε λοιπόν πρώτα την προστιθέμενη αξία ενός ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης ανεργίας. Το θέμα είναι λοιπόν ότι η μακροπρόθεσμα μακροοικονομικά θα μπορούσε να λύσει ένα πρόβλημα συντονισμού. Το πρόβλημα είναι για τις μικρές οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι σε περίπτωση δημοσιονομικών κλονισμών ε, ε, κάθε κράτος ε, έχει περιορισμένη δυνατότητα αντίδρασης επειδή οι συνέπειες περνάνε και σε άλλες οικονομίες. Εάν λοιπόν ο καθένας ε, φερθεί λογικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε μια αντίδραση μη ιδανική. Αυτό μπορεί να λυθεί αν έχουμε κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά θέλουμε ε, να αρθούν οι περιορισμοί ε, στην ανταπόκριση απέναντι στην ευρωπαϊκή κρίση. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούν να ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό λοιπόν θα μπορούσε να λύσει το περιορισμένο πεδίο κίνηση ε, των ε, εθνικών κυβερνήσεων και επίσης ε, θέλουμε να διευκολύνουμε την διασυνοριακή κινητικότητα των εργαζομένων. Έχουμε προσθέσει και το πολιτικό σκεπτικό, αλλά αυτό βέβαια είναι μάλλον κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσετε εσείς. Θα μπορούμε σε πολιτικό επίπεδο όμως να ανταποκριθούμε στο αίτημα των πολιτών για πιο κοινωνική Ευρώπη. Τέσσερις προσωμιώσεις κάναμε. Να σας παρουσιάσω λοιπόν σύντομα. Δύο μοντέλα συγκρίναμε. Το ένα είναι το εναρμονισμένο επίδομα ενέργειας Συλλέγονται δηλαδή τα χρήματα από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο κάθε χρόνο στέλνει σε κάθε κράτος ε, τα επιδόματα που χρειάζεται. Αυτό λοιπόν αποτελεί μερική αντικατάσταση των εθνικών συστημάτων από το ευρωπαϊκό σύστημα. Η Ευρώπη λοιπόν εγγυάται ότι κάθε ε, Ευρωπαίος πολίτης ε, θα λάβει τέτοιο επίδομα. Ένα καταστροφικό επίδομα έχει διαφορετική φύση, έτσι το ονομάζουμε, ουσιαστικά θα πληρώνονται χρήματα μόνο σε, ε, στις εθνικές κυβερνήσεις σε περίπτωση σημαντικών ε, αναταραχών, ε, σε, σημαντικών κλειδονισμών στην οικονομία. Σε τέτοια περίπτωση λοιπόν θα παρέχει δημοσιονομικούς πόρους ε, στις εθνικές κυβερνήσεις για να μπορέσουν να συμπληρώσουν το σύστημα ανεργίας. Γι' αυτό το ονομάζουμε καταστροφικό, δηλαδή για περίπτωση καταστροφής. Επίση, η προσωμείωσή μα εξετάζει δύο περιπτώσεις ε, όσον αφορά τον προπολογισμό. Η βασική λύση είναι τα συστήματα αυτά να λειτουργούν όπως σας εξήγησα σύντομα, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις ε, αυτό θα οδηγήσει σε μακροπρόθεσμες μεταφορές εισοδήματος από ένα κράτος μέλος σε κάποιο άλλο. Διότι κάποια κρατημέλη έχουν προβλήματα πιο σοβαρά από άλλα. Ακόμα και αν λάβουμε υπόψη μας ε, την μόνιμη ανεργία και την διαρθρωτική ανεργία. Ε, ε, εμπνευσμένοι εν μέρει από τι Ηνωμένε Πολιτείε, ε, προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε μία λύση ουδέτερη ω προς τον προϋπολογισμό. Θα σας εξηγήσω λοιπόν πώς το σχεδιάσαμε αυτό. Θέλουμε λοιπόν στην λύση Β να φροντίσουμε κανένα κράτος μέλος να μην φτάσει σε σημαντικά ελλείμματα. Κάποια στιγμή δηλαδή υπάρχει ένα φρένο με μεταφορών εισοδήματος προς κάποια συγκεκριμένη χώρα. Κοιτάξαμε αναδρομικά το διάστημα από το 1991 μέχρι το 2012. Ε, επιλέξαμε αυτές τις ημερομηνίες επειδή τίθεται αφενός θέμα διαθεσιμότητας δεδομένων ε, για τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ε, και συμβολικό διότι το 1999 είναι η έναρξη της τελευταίας φάσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, δηλαδή της πραγματικής δημιουργίας της Ευρωζώνης, της πρακτικής δημιουργίας Ευρωζώνης. Το θέμα λοιπόν είναι Ε, τι συμβαίνει μετά το 1999 είναι απλή η προσημείωσή μας. Ε, δεν μπορέσαμε να λάβουμε υπόψη μας σε κάποια δευτερογενή οικονομικά αποτελέσματα, διότι έτσι θα είχαμε πολύ, ε, πλοκό οικονομικό μοντέλο, αλλά για κάποιου λόγου δεν θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερο πολύτιμα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι έχουμε καλύψει τα βασικά. Επιτρέψτε μου τώρα να εξηγήσω πιο αναλυτικά τις δύο προτάσεις. Η πρώτη για την εναρμονισμένη ασφάλιση ανεργίας Ε, προβλέπει ότι το 75% των εργαζομένων ε, που είναι άνεργοι για λιγότερο από ένα χρόνο θα καλυφθούν. Ε, αν το συγκρίνετε αυτό με τα νούμερα στην έκθεσή μας, θα διαπιστώσετε ότι είναι υψηλότερο το νούμερο αυτό από την κατάσταση σε περισσότερες, στις περισσότερες χώρες. Τα περισσότερα κρατημέλη έχουν χαμηλότερη κάλυψη. καλύπτεται το 25%. Είναι δηλαδή πιο ολοκληρωμένο το δικό μας σύστημα από τα περισσότερα εθνικά συστήματα το 40% της, ε, της αποζημίωσης τους ακαλύπτει, ε, το σύνολο δηλαδή του εργασιακού κόστους, ε, όχι μόνο του μισθού. Διότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συγκρίνουμε πιο εύκολα. Και θα πληρώνεται αυτό το επίδομα για 6 μήνες κατά μέσο όρο. Προβλέπουμε λοιπόν ε, έναν φόρο 0,5% της συνολικής αποζημίωσης ε, άσχετα από το αν το πληρώνει αυτό ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος. Η ασφάλεια σε περίπτωση καταστροφής ε, έχει περίπου παρόμοια επίπεδα γενεοδορίας αλλά έχει διαφορετικό σημείο κινητοποίησης. Εάν το ποσοστό ανεργίας ε, σε μια χώρα ξεπεράσει τον Ναύρου που είναι η μόνιμη ανεργία, η μακροπρόθεσμη ανεργία, εάν δηλαδή αυτό το ποσοστό φτάσει πάνω από 2% ε, στέλνει το Ταμείο αυτό χρήματα στις εθνικές κυβερνήσεις. Αποστέλλονται χρήματα κατά τα άλλα, όπως ε, και στο Ευρωπαϊκό ενερμονισμένο Σύστημα Ασφάλισης Ανεργίας. Αλλά τα ε, ο φόρος είναι πολύ πιο χαμηλός διότι ε, δεν είναι μόνιμο το σύστημα αυτό, ή είναι μόνο σε περίπτωση καταστροφής. Κάθε κράτος μέλος λοιπόν ε, χρειάζεται να συνεισφέρει με το 0,1% του ΑΕΠ του κάθε χρόνο μέχρι να συμπληρωθεί το Ταμείο και κατόπιν σταματάνε οι, οι συνεισφορές εφόσον ε, δεν πέφτει κάτω από 0,5% του ΑΕΠ ε, το ταμείο. Εδώ λοιπόν βλέπετε κάποια διαγράμματα. Εάν ε, δούμε τις ετήσιες δαπάνες βλέπετε αμέσως τη διαφορά ανάμεσα στα δύο συστήματα. Η μπλε γραμμή, η πάνω γραμμή είναι το εναρμονισμένο σύστημα το οποίο εν μέρει αντικαθιστά τα εθνικά. Στοιχίζει πολύ περισσότερο διότι στέλνει χρήματα για κάθε άνεργο 0,25 με 30% στις ε, καλές ε, εποχές ε, φτάνει μέχρι 40% σε περίοδους κρίσης. Ενώ το άλλο βλέπετε ότι βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Σε καλές εποχές η συνεισφορά είναι γύρω στο 0 μάλλον τα χρήματα που αποστέλλονται προς τα κράτη-μέλη είναι πολύ χαμηλά. Ε, σε περίπτωση κρίσης ε, αυξάνεται πολύ. Παρ' όλα αυτά ε, παραμένει πολύ πιο χαμηλά όσον αφορά το ποσοστό του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Στο επόμενο σχέδιο βλέπετε την σε, εθνικό, σε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι γίνεται. Το, το σύστημα καταστροφής λοιπόν ε, έχει πολύ πιο υψηλό σημείο ισορροπίας. Ε, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά βέβαια είναι πολύ πιο εύκολο αν έχουμε συγκεντρώσει κάποιο ταμείο για δύσκολες εποχές από ότι εάν ζητάμε από τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν στους δύσκολους καιρούς. Το εναρμονισμένο σύστημα Ε, συσσωρεύει πολύ λιγότερα. Εάν κοιτάξετε τις αιτήσιες ε, ισορροπίες βλέπετε ότι σε καλές εποχές έχουμε κάποιο μικρό πλεόνασμα, σε κακές εποχές έχουμε ένα μικρό έλλειμμα, αλλά πολύ ελαφρά είναι αντισυγκυριακό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ σε εθνικό επίπεδο η εικόνα είναι πολύ διαφορετική. Και αυτό φαίνεται στην επόμενη διαφάνεια, όπου Βλέπουμε τη δυνατότητα σταθεροποίηση. Βλέπετε εδώ πέρα το ποσοστό ΑΕΠ που αποστέλλεται στα κράτη-μέλη συνολικά μέσα σε 14 χρόνια. Βλέπετε λοιπόν τις συνεισφορές τους, μείον αυτά που έλαβαν. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι για τις χώρες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση η ασφάλεια σε περίπτωση καταστροφής προβλέπει πολύ εκτενή ε, κάλυψη. Για την Ισπανία βλέπουμε το 4% του ΑΕΠ, αλλά ακόμα και για τις χώρες της ε, Βαλτικής εκειμένεται από 1 2% ε, του ΑΕΠ. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό ισχύει όμως και για κάποιες χώρες της Νότιας Ευρώπης. Παρά λοιπόν το μικρό του μέγεθος σε δύσκολους καιρούς μπορεί να παράσχει βοήθεια αυτού του είδους η ασφάλιση. Ε, δεν έχω πολύ χρόνο, θα σας δώσω όμως δύο παραδείγματα. Έχουμε την ε, Λετωνία που είναι ένα υπόδειγμα του πώς θα πρέπει να λειτουργεί το σύστημα αυτό. Βλέπετε τον ετήσιο ισολογισμό για την ε, Λετωνία και στις δύο περιπτώσεις. Βλέπουμε ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης έχουμε πολύ αρνητικά νούμερα διότι η Λετωνία επλήγει σημαντικά από την κρίση Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα ένα αντικυκλικό κίνητρο, αντισυγκυριακό κίνητρο. Ε, βλέπουμε όμως και μία ανάκαμψη για λόγους που θα σας εξηγήσω σε λίγο. Η Ισπανία αποτελεί άλλη ενδιαφέρουσα περίπτωση. Είναι μια από τις χώρες που θα υποφελθούν περισσότερο από το σύστημα αυτό κατά ε, τις περιόδους ε, κρίσης. όταν ξεκινάει λοιπόν η κρίση και στις δύο περιπτώσεις η Ισπανία έχει πολύ σημαντικό έλλειμμα στο σύστημα αυτό. Υπάρχουν πολλές περισσότερες ε, μελέτες σε συγκεκριμένων περιπτώσεων. Έχουμε δώσει νούμερα ε, των χωρών που θα είναι συνεισφορή, σε ποιες χώρες ε, θα αλλάζουν ρόλο κατά καιρούς, αλλά οι περισσότερες χώρες μπορούν μακροπρόθεσμα να είναι κοντά στο μηδέν. Για κάποιες χώρες όμως αυτό θα είναι δύσκολο. Για παράδειγμα ήταν δύσκολο να σχεδιάσουμε ένα σύστημα όπου η Αυστρία και οι κάτω χώρες να μην είναι καθαροί ε, ε, συνεισφορείς, διότι δεν ε, έχουν υποστεί καμία κρίση τα τελευταία 14 χρόνια και επίσης θα ήταν δύσκολο να βρούμε ένα σύστημα όπου δεν θα υποφελείται η Ισπανία επειδή είχε τόσο σημαντική ανεργία στο παρελθόν. Αυτό βέβαια δεν αποδεικνύει τίποτα για το μέλλον. Ε, μπορεί σε πέντε χρόνια να έχουμε δύσκολη κατάσταση στην ε, Αυστρία και να είναι πολύ διαφορετικά τα νούμερα από ό,τι στο παρελθόν. Ε, θα πηρήξω τη διαφάνεια αυτή, δεν είναι τόσο σημαντική και θα περάσω στην επόμενη. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε μόνιμες ε, μεταφορές πόρων. Στην λύση Β, λοιπόν, δείχνουμε πώς μπορούμε να μειώσουμε τις μόνιμες ε, μεταφορές ε, πόρων ε, με ένα πολυσύστημο σύστημα. Όταν το συγκεντρωτικό έλλειμμα μιας χώρας ξεπερνάει το 1% του ΑΕΠ, όταν δηλαδή έχει λάβει ε, ε, ε, περισσότερο από αυτό το ποσοστό από ό,τι έχει πληρώσει, θα πρέπει να συνεχίσει να συνεισφέρει περισσότερα. Συνεχίζει δηλαδή να λαμβάνει πόρου, αλλά θα πρέπει να συνεισφέρει επίση ή να εξισορρεπήσει την συνεισφορά του. Έχουμε εμπνευστεί από τι ΗΠΑ για το θέμα αυτό. Στη φύση του μοιάζει πολύ με το σύστημα τη Αμερική. Ουσιαστικά δηλαδή δεν είναι μηχανισμός μεταφορά εισοδήματος αλλά σύστημα απορρόφηση των κραδασμών. Έχουμε λοιπόν τη λύση Α που δεν υπάρχει αυτό και τη λύση Β όπου προτείνεται ακριβώ ε, αυτό. Μπορείτε λοιπόν εσεί να κοιτάξετε τι δύο λύσει και να επιλέξετε ποια προτιμάτε. Και προχωρώ τώρα στα συμπεράσματα πολύ σύντομα. Τη μελέτη μας ε, τη βασίσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο στην Ευρωζώνη. Ε, γιατί, διότι κάποιες χώρες έτσι σταθεροποιούν περισσότερο το σύστημα, αλλά επίσης δεδομένης της αύξηση της Ευρωζώνης, βλέπουμε την Εστονία, τη Λετονία, την ε, Λιθουανία, ε, βλέπουμε ότι, ο, η, η, ότι η Ευρωζώνη είναι κινούμενος στόχος, γι' αυτό επιλέξαμε να εξετάσουμε το σύλλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντως παρόμοια μορφή θα έχει το σύστημα αν εξετάζαμε μόνο την Ευρωζώνη. Δύο μεγάλες οικονομίες ε, βρίσκονται εκτός Ευρωζώνης, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Πολωνία. Η Πολωνία έχει πιο χαμηλό κατακεφαλήν ΑΕΠ, έτσι δεν ε, συνεισφέρει τόσο σημαντικά ε, στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά λοιπόν ε, το Ηνωμένο Βασίλειο κάνει τη διαφορά, αλλά δεν θα άλλαζε ούτε και αυτό σημαντικά την εικόνα. Προτείνουμε υποχρεωτική συμμετοχή, ώστε να μην μπορούν να επιλέξουν τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν. Έχει λοιπόν ε, νόημα να υιοθετήσει ή να μην υιοθετήσει κανεί το σύστημα, όχι όμω να το προσφέρει ω επιλογή στα κράτη-μέλη. Όσον αφορά του δείχτε, προτείνουμε. Την ε, διαφορά στα, στα ποσοστά ανεργία, δηλαδή ανάμεσα στη μακροπρόθεσμη και την ε, βραχυπρόθεσμη ανεργία, το πόσοι δεν έχουν δουλειά ε, πάνω από ένα χρόνο και κάτω από ένα χρόνο. Ε, έτσι, ουσιαστικά μηδενίζουμε τι τις συνέπειε τη της διαθροτικής ανεργίας. Η, η Ισπανία ή η Σλοβακία έχουν πολύ ψηλότερη μακροπρόθεσμη ανεργία από ότι η Γερμανία ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλουμε να απορροφούνται οι κρατασμοί και γι' αυτό επιλέγουμε τους κατάλληλους δείκτες. Το άλλο θέμα είναι η εξισορρόπηση του ε, οικονομικού κύκλου, της οικονομικής συγκυρίας. Ήδη σας εξήγησα ότι προσπαθήσαμε να περιορίσουμε το όφελος ε, των χωρών ε, στο 1% του ΑΕΠ μακροπρόθεσμα. Εάν δεν είχαμε ένα τέτοιο σύστημα, δεν θα άλλαζαν πολλά συνολικά. Δηλαδή, αν κοιτάξετε το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν υπάρχει αυτό το όριο του 1% του ΑΕΠ, αυτό δεν αλλάζει πολλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλάζει όμως σε επίπεδο κρατών μελών. Η Ισπανία θα επωφελεί το πολύ περισσότερο εάν ε, δεν υπήρχε το όριο αυτό. Είναι λοιπόν πολιτικό το σύστημα, θέλουμε να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο ή όχι. Μας ενδιαφέρει άλλωστε η δημοσιονομική σταθερότητα και στην ε, τελευταία διαφάνεια των συμπερασμάτων ε, βλέπετε όσον αφορά τη φορολογία. Για το εναρμονισμένο σύστημα προβλέπουμε να χρηματοδοτείται με την ε, φορολογία εισοδήματος. Γι' αυτό προτείνουμε το 0,5% της ε, ονομαστικής αποζημίωσης. Η ασφάλιση καταστροφών ε, δεν έχει να κάνει με τη σχέση του ατόμου με το σύστημα. Είναι χρήματα που δίδονται στο κράτος μέλος, οπότε προτείνουμε ε, συνεισφορά του κράτους όσον αφορά το μέγεθος αυτής, αυτό υπολογίζεται διαφορετικά. Η τελευταία παρατήρηση που θέλω να κάνω έχει να κάνει με το ερώτημα που μας έθεσαν. Θα πρέπει να υπάρχουν κοινά πρότυπα για την ε, ευρωπαϊκή ασφάλιση ανεργίας. Αυτό απαντάται με τον εναρμοσμένο σύστημα, διότι έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει τους κανόνες ε, προς ε, τα κράτη-μέλη για την ε, πληρωμή των επιδομάτων ενεργείας. Κάθε πολίτης δηλαδή που πληρεί τα εξής κριτήρια θα δικαιούται την, το επίδομα ενεργείας. Πολιτικά μπορεί να καθοριστεί το επίπεδο εναρμόνισης, ε, αλλά αυτό ε, είναι πολύ περισσότερο από ό,τι ισχύει για το σύστημα ασφάλισης σε περίπτωση καταστροφής. Διότι ε, αυτό, σε αυτό ισχύει ότι λέμε, ωραία, μια χώρα συναντάει προβλήματα, της δίνουμε τα χρήματα, Εκεί δεν χρειάζεται να πούμε στο κράτος μέλος πώς θα ξοδέψει τα χρήματα. Θα μπορούσε όμως να περιγράψει κανεί και πάρα πολύ αναλυτικά πώς θα πρέπει το κράτος μέλος αυτό να δαπανίσει τα χρήματα. Πρόκειται για πολιτική επιλογή. Η δική μας ε, σύσταση, αλλά πολύ επιφυλακτικά, είναι να υπάρχει να υπάρχουν μερικές προϋποθέσεις, δηλαδή ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, τα χρήματα αυτά για επίδομα ανεργίας ε, για να ε, έχουμε ένα αντικυκλικό αποτέλεσμα, αλλά να μην περιορίσουμε τη διακριτική ευκαιρία των κρατών μελών στο θέμα αυτό. Αυτά από εμά. Ε, προσπάθησα να είμαι σύντομο, ξέρω ότι σε πέρασε το χρόνο μου, θα σταματήσω εδώ και είμαι στη διάθεσή σα να απαντήσω σε ερωτήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ. Α δούμε την παρουσίαση τη άλλη μελέτη. για να υποβάλουμε ερωτήσεις στη συνέχεια. Η δεύτερη μελέτη διενεργήθηκε από το, ε, το Centrum für Europäische Wirtschaftsforschung της Γερμανίας και το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβέν. Έχετε το λόγο για 15 λεπτά επίσης. Ευχαριστώ και θα ήθελα να ζητήσω, να σας ευχαριστήσω γιατί μας δίνετε την δυνατότητα να πλησιάσουμε το σχέδιό μας ε, μέσα στα πλαίσια ενός προγράμματος ε, καταπολέμησης της ανεργίας. Θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω αυτά στοιχεία που αφορούν την προστασία του εισοδήματος με βάση τους οργανισμούς αντιμετώπισης ανεργίας. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να ξέρουμε κάτι για την προστιθέμενη αξία ε, ενός ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης. Άρα θα πρέπει να δούμε καταρχήν τα εθνικά. Στη συνέχεια θα μιλήσω για τα ε, χαρακτηριστικά του συστήματος ασφάλισης της Ευρωζώνης και Ευρωζώνης και θα μιλήσω και για τα συστήματα όπως έχουν εξελιχθεί. Δηλαδή θα επικεντρωθούμε στην Ευρωζώνη γιατί οι μηχανισμοί είναι οι ίδιοι για την Ευρωζώνη και μετά στο κυρίως τμήμα θα μιλήσω για τις προσωμιώσεις που διενεργούνται και τα βασικά αποτελέσματα. Νομίζω ότι η προστιθέμενη αξία της ε, μελέτης μας είναι ότι χρησιμοποιούμε ε, μακροδεδομένα σε σχέση με τα νοικοκυριά και στην χώρα και σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί έχουμε εμπειρικά στοιχεία στα νοικοκυριά όπου υπάρχουν μεγάλες ε, διαφορές σε σχέση με τα ε, διάφορα ε, στοιχεία κατανάλωσης ή σχήματα κατανάλωσης. Και τέλος, θα σας μιλήσω για τα βασικά συμπεράσματα. Σε σχέση με την ε, προστασία εισοδήματος από τα εθνικά συστήματα ασφάλισης πριν από την κρίση, εδώ έχω στοιχεία από προγενέστερες μελέτες όπου προσωμιώσαμε τους κλειδονισμούς ανεργίας στις χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, ε, πρόκειται για ένα πείραμα όπου αυξήσαμε κατά 5% το δίκτυ ανεργίας. Πρόκειται για ένα υποθετικό σενάριο κλειδονισμών με βάση τις εθνικές παραμέτρους και τα μικροδεδομένα πριν από την έναρξη της κρίσης και βλέπουμε τον συντελεστή σταθεροποίησης εισοδήματος για να δούμε κατά πόσο οι κλειδονισμοί αντιμετωπίζονται. Βλέπουμε ποιες είναι οι δυνατότητες απορρόφησης αυτών των κλειδονισμών. Πριν από την κρίση βλέπουμε ότι ένα 25% αυτών των κλειδονισμών απορροφάται και υπάρχει και σταθεροποίηση στις ανατολικές και νότιες χώρες της Ευρώπης. Υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι, υπάρχουν ε, διαφορετικοί βαθμοί γενεοδορίας, άλλοι όροι εκλογιμότητας των ανέργων έτσι ώστε να τους ε, καταβληθεί το επίδομα. Και γι' αυτό βρίσκουμε διαφορετικά επίπεδα προστασίας του εισοδήματος. Επίσης, τεκμηριώνουμε στην έκθεσή μας τα σχέδια αυτά και τα σχήματα αυτά που ε, άλλαξαν κατά τη διάρκεια της ε, κρίσης. Ε, δηλαδή, οι χώρες που έχουν χαμηλή σταθεροποίηση ε, τόνισαν την ε, σταθεροποίηση αυτή με βάση νέες πολιτικές. Τα υπάρχοντα αποδεικτικά στοιχεία δεν καταδεικνύουν ότι υπάρχει πραγματική η σταθερότητα στα εθνικά συστήματα ασφάλισης. Τώρα, τα, ως προς τα βασικά ή τα ενδυνάμει χαρακτηριστικά της Ευρωζώνης, εδώ θα είμαι πολύ σύντομος, διότι ο συνάδελφος μίλησε για τις ενελεκτικές και αυτά τα στοιχεία που δώσαμε, η πρώτη εναλλακτική είναι ένα βασικό σχέδιο σχήμα ε, αντιμετώπισης ανεργίας. Δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ελάχιστο επίπεδο ε, ασφάλισης, σε ένα 50% για 12 μήνες. Αυτή θα είναι η κάλυψη και μετά τα εθνικά συστήματα θα μπορούσαν να ε, προσθέσουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό αν το ε, επιθυμούν. Βεβαίως η γενεοδορία διαφέρει από κράτος σε κράτος. Η δεύτερη εναλλακτική θα ήταν μια ε, επέκταση του προγράμματος ευεργετημάτων όπως ισχύει στο, στις ΗΠΑ ανάλογα με τα επίπεδα ανεργίας ή τις αλλαγές για τις καταβολές αυτές. Αυτό το σύστημα θα ήταν συμπληρωματικό στα εθνικά, δίνοντας επιπλέον επιδόματα. Και το τρίτο και η τρίτη εναλλακτική θα ήταν να υπάρχει ένα σύστημα, ευρωπαϊκό σύστημα αντιμετώπισης ανεργίας, το οποίο θα αντικαταστήσει τα εθνικά. Ε, και θα σήμαινε ότι τα εθνικά συστήματα καταργούνται. Εδώ ε, θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να προγραμματιστεί ένα τέτοιο σύστημα με βάση τα προϋπάρχοντα και κατά πόσο θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε έναν μέσο όρο τρία συστήματα έχουν διαφορετικές ε, επιπτώσεις ανάλογα με τα κίνητρα που προσδίδονται από την νέα κατανομή αλλά και την ε, διοικητική χειραγώγηση. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, πιστεύω όμως ότι ε, έχετε όλα τα στοιχεία στην έκθεσή μας. Ως προς την εμπειρική ανάλυση, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ένα σύστημα ασφάλισης και καταπολέμηση της ανεργίας. Χρησιμοποιούμε μικροστοιχεία, δηλαδή με βάση τον υπολογισμό Euromod και χρησιμοποιούμε στοιχεία προκρίσης το 2007, διότι δεν έχουμε στοιχεία για την Ευρωζώνη των 17 και μετά έχουμε διασταυρούμενες μελέτες για την περίοδο 2008-2013. Δηλαδή χρησιμοποιούμε το στοιχείο της Euromod που επιτρέπει προσωμιώσεις. Επίσης, η ανάλυση μας δείχνει τι θα είχε συμβεί αν υπήρχε ένα κοινό ε, σχέδιο ή πρόγραμμα ασφάλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της προσομοίωσης αυτής και του συστήματος ασφάλισης θα είχαμε ένα σύστημα αντικατάστασης κατά 50% και θα είχαμε τέτοια κάλυψη έτσι ώστε να είναι ένα ουδέτερο σχήμα για την περίοδο 2008-2013. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ελλείμματα και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει σταθεροποίηση με βάση μία απτή χρηματοδότηση έτσι ώστε να μην υπάρχει αποσταθεροποίηση σε μεγάλη κρίση σε ολόκληρο το επίπεδο της Ευρωζώνης, διότι διαφορετικά οι χώρες που δεν θα είχαν πληγεί τόσο θα αποσταθεροποιηθούν. Θα μπορούσαν να αποσταθεροποιηθούν τα μικροστοιχεία. Μας επιτρέπουν να δούμε τον αριθμό ανέργων που θα ήταν επιλέξιμοι για το πρόγραμμα αυτό, διότι ξέρουμε ποιοι είναι άνεργοι βράχοι πρόθεσμα ή άνεργοι που είχαν προγενέστερη απασχόληση. Έχουμε λοιπόν μία σχεδόν πλήρη κάλυψη, δηλαδή καλύπτουμε περίπου το 50% των ανέργων. Ο προϋπολογισμός θα ήταν 365 δις ευρώ για την περίοδο 2008 2013, άρα θα είχαμε 61 δις ευρώ ετησίως. Εδώ βλέπετε την εξέλιξη των δικτών ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη δηλαδή, για τη Γερμανία και τις χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση και βλέπουμε ξεκινώντας από το 2001 ότι υπάρχουν διάφορες υποπερίοδοι. Το 2005 ας πούμε η Γερμανία είχε ένα δίκτυο ανεργίας που θα μπορούσε να είναι συγκρίσιμος ε, με άλλες χώρες και ήταν χαμηλός και στις ε, χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει μόνιμη αναδιανομή καθε αυτή. Όλα εξαρτώνται από την ε, αλλαγή, τις αλλαγές της, ε, βραχυ, της βραχυπρόθεσμης ανεργίας. Το 2007 βλέπουμε μια μεγάλη απόκληση η Γερμανία ακολουθεί ευθύνουσα πορεία και στην Ελλάδα και Ισπανία είχαμε ένα 27-30% δίκτυα ανεργίας. Τώρα ως προς το δίκτυο κάλυψης το βασικό μήνυμα από αυτή τη γραφική παράσταση είναι ότι ένα βασικό σχήμα ασφάλισης που καλύπτει τους δύο τους πρώτους 12 μήνες εξαρτάται από τη βραχυπρόθεσμη ανεργία. Και βλέπουμε εδώ ότι έχουμε ένα μειούμενο δίκτυ κάλυψης. Άρα το 2009 στην αύξηση της ανεργίας υπήρχε κάλυψη, αλλά τα επόμενα χρόνια επειδή αυξήθηκε η μακροχρόνια ανεργία δεν μπορούσε να υπάρξει πλήρης κάλυψη, άρα δεν υπήρχε ε, εκλογιμότητα εδώ. Άρα ένα βασικό ε, πρόγραμμα ασφάλισης ασφαλίζει τους ανέργους για μια βραχυχρόνια περίοδο, αλλά όχι μακροχρόνια. Στην Ισπανία βλέπουμε ότι έχουμε δείκτη κάλυψη 67% το 2008, αλλά έπεσε σε 52% το 2013 και στην Ελλάδα ο δείκτης κάλυψης έπεσε από το 53% το 2008 σε 38% το 2013. Βλέπετε επίσης τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο όπου έχουμε μειούμενο ε, δείκτη και ένα ε, βασικό, μια φθήνουσα πορεία μέσα στα πλαίσια της προσωμείωσης. Τι γίνεται ως προς τις καθαρές εισφορές στις χώρες. Θα το δούμε σε επίπεδο ευρωζώνης καταρχήν. Θα είχαμε πλεονάσματα καταρχήν ε, τα 2008, 10 και 11 και ελλείμματα το 10, ε, 11 και 13. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό δεν ισχύει σε κρατικό επίπεδο. Βλέπουμε ότι οι μεγαλύτεροι θα ήταν η Αυστρία, η Γερμανία και το Βέλγιο και η Ολλανδία και η Ισπανία, η Γαλλία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία θα ήταν οι μεγαλύτεροι οφειλέτες. Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος εισφορέας 7,4 έως 13 δις ευρώ. Τέλος, πώς ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να οδηγήσει σε σταθεροποίηση, ποια είναι η προστιθέμενη αξία αυτού του σχεδίου. Είπα στην αρχή ότι η χώρες, οι ορισμένα κράτη-μέλη δεν θα μπορέσουν να ε, ε, επιφέρουν σταθεροποίηση διότι δεν υπάρχουν δεν υπάρχουν πιστώσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μια κυκλική ε, φορολογική πολιτική σε περίοδο κρίσης. Σε επίπεδο χρηματοδότησης λοιπόν θα μπορούσαμε να έχουμε χαμηλότερες εισφορές και υψηλότερα ευεργετήματα. Άρα εδώ βλέπουμε πώς ένα ευρωπαϊκό σχέδιο θα μπορούσε να βοηθήσει στη σταθεροποίηση για τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερα. Βλέπουμε ότι το βασικό στοιχείο αφορά αυτές τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερα, αλλά το 2009 η Ευρωζώνη θα είχε ένα δίκτυ σταθεροποίησης ακόμη. Κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει με ένα σχέδιο χρηματοδότησης του χρέους. Όπως βλέπετε την φθήνουσα πορεία κάλυψης, βλέπουμε ότι ε, το 2009 είχαμε ένα 50% στην Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία, αλλά η σταθεροποίηση ακολουθεί πτωτική πορεία διότι η ανεργία γίνεται μακροχρόνια. Η Ελλάδα και η Ισπανία είναι οι μόνες χώρες που θα μπορούσαν να είναι σταθεροποιημένες κατά την περίοδο προσωμίησης το οποίο σημαίνει ότι αυτό το σχέδιο ε, καλύπτει τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. Τέλος, ε, στα συμπεράσματα ξέρω ότι δεν έχω πολύ χρόνο. Θα ήθελα να πω ότι ένα βασικό στοιχείο είναι ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια πλήρη κάλυψη με χαμηλό προϋπολογισμό, δηλαδή 61 δις το 2008-2013, που ήταν μια έκτακτη περίοδος. Πριν το 2008 αυτό το σύστημα ασφάλισης θα είχε χαμηλότερο προϋπολογισμό. Και το πλεονέκτημα είναι ότι δεν υπάρχει επανακατανομή εξ άντε. Όμως, υπάρχει και ε, μεγαλύτερος κίνδυνος διοικητικών ε, χειραγωγήσεων και μοχλεύσεων, δηλαδή επιδότηση των ε, μισθών. Άρα οι άνεργοι θα μπορούσαν που δεν είναι επιλέξιμοι θα μπορούσαν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή τη δυνατότητα μόχλευσης. Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο αναμονής ή απασχόλησης πριν από τη χορήγηση επιδόματος. Όσο μεγαλύτερες είναι οι περίοδοι αυτοί, τότε θα ήταν και πιο δαπανηρό το σχέδιο και θα μπορούσε να τύχει μόχλευσης. Όμως ε, θα είχαν μεγαλύτερα αποτελέσματα και τα σχέδια ασφάλισης αυτά. Τι θα μπορούσε, πώς θα μπορούσαμε να δράσουμε σε επίπεδο σταθεροποίησης μέσα στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού συστήματος αντιμετώπισης ανεργίας. Νομίζω ότι μακροχρόνια θα υπήρχε ε, μία μετριοπαθής ε, εξέλιξη. Όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να τα δούμε μακροχρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ και τους ε, δύο, γιατί βεβαίως και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για ομαδικές προσπάθειες. ξεκαθαρίσετε πολλά ζητήματα που μας απασχολούν. Όπως ξέρατε, ξεκινήσαμε και με μια ακρόαση ε, στην Επιτροπή μας πριν από ένα χρόνο περίπου. Με εξέπληξε που στη δεύτερη μελέτη θεωρείται ότι οι μακροοικονομικές επιπτώσεις ε, έχουν αντίκτυπο μόνο το πρώτο έτος, από ό,τι κατάλαβα. Πρέπει να δούμε και από την ε, πρώτη μελέτη τους εκπροσώπους αν συμμερίζονται αυτή την ε, εκτίμηση. Γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό σημείο στην επιχειρηματολογία σε ό,τι αφορά την προστιθέμενη εξέτου συστήματος. Στη δεύτερη μελέτη, μεταξύ του πρώτου γραφήματος ε, που εντοπίζει τα εφιστάμενα συστήματα και τον τρόπο με τον οποίο θα είχαμε μια κάλυψη ανά κράτος μέλος με αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα, δεν βλέπουμε ακριβώς την ίδια καμπύλη. Τι σημαίνει λοιπόν στο μεταξύ, εφόσον δεν υπάρχει αναρμόνιση όλων των όρων ε, επιδομάτων και των διαφορετικών τρόπων επιδότησης, πώς, για παράδειγμα, στο Λουξεμβούργο η κάλυψη είναι τόσο χαμηλή. Α, γιατί στη μία περίπτωση μιλούμε για το ποσό, στην άλλη μιλάμε για το ποσοστό. Α, το ποσοστό της κάλυψης. Ίσως είναι αυτή η δυσκολία. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια σύγκριση. Πώς αυξάνεται ή όχι το ποσοστό κάλυψης ε, με βάση τα εφιστάμενα συστήματα. Και αν δείτε το θέμα των καθαρών εισφορών, θέλω και πάλι να δω αν υπάρχει ε, κοινή αντίληψη μεταξύ των δύο μελετών για τα ωφέλη αυτού του συστήματος. Πριν σας δώσω και πάλι το λόγο, να δω αν κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Σρέντερ. Ναι, καταρχάς να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις μελέτες, είναι πολύ σημαντικές. Γίνεται μεγάλη συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό, αν θα πρέπει να το κάνουμε ή όχι. Κάποιοι θεωρούν μάλιστα ότι πρέπει να τροποποιηθεί η συνθήκη, αν θέλουμε να εισάγουμε τέτοια συστήματα. Γι' αυτό έχω δύο ερωτήσεις. Η μία ερώτηση είναι πόσο θα πρέπει να περιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή πόσο δεν θα πρέπει να περιμένει για να εισάγει το σύστημα. Αυτή τη στιγμή περνάμε μια κρίση. Με το σύστημα αυτό δεν μπορούμε πια να αντιδράσουμε. Διότι θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να εισαχθεί ένα τέτοιο σύστημα. Πιθανότατα σε 5-6 χρόνια, όταν θα μπορέσουμε να έχουν διαμορφωθεί πολιτικά τέτοια συστήματα, θα μπορούσαμε να το έχουμε. Εσείς έχετε κάποια χρονική διάσταση, δηλαδή αν η Ευρωπαϊκή Ένωση πει δεν κάνουμε τίποτα τώρα, περιμένουμε 10 χρόνια, αυτό μπορεί να έχει μειονεκτήματα. Πόσο μάλλον που άλλες μεγάλες οικονομίες έχουν ένα τέτοιο σύστημα. Αυτή είναι η μία ερώτηση και η δεύτερη είναι... Από ό,τι κατάλαβα από την πρώτη παρουσίαση, αυτό το βασικό επίδομα ανεργίας ε, είναι το μόνο καλό σύστημα, διότι υπάρχει σχετικά γρήγορα ε, εξισορρόπηση και δεν είναι τόσο μεγάλο το κόστος. Εγώ θα ήθελα να γνωρίζω, εσείς πόσο χρόνο πιστεύετε ότι χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εισάγει ένα τέτοιο σύστημα, από την πολιτική απόφαση δηλαδή, μέχρι να λειτουργήσει στην πράξη. Μέχρι να δούμε δηλαδή τα οικονομικά αποτελέσματα. Πόσο θα διαρκέσει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω ποιος έλει να μιλήσει πρώτος. Σέψ πρώτα. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω και μετά θα πάρει το λόγο ο συνάδελφο για να συμπληρώσει. Ε, σε τρία τίγματα θα απαντήσω. Πρώτον, για την αποτελεσματικότητα ε, στο πρώτο έτος ε, του κλειδονισμού σε σχέση με τις πιο μακροχρόνιες επιπτώσεις τα επόμενα έτη. Επί της αρχής και τα δύο αυτά σχήματα αφορούν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Δεν υπάρχει λοιπόν για μα διάκριση μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου έτου. Όμως υπάρχουν δύο παράγοντες που μειώνουν τον αντίκτυπο ε, με τον καιρό. Μπορούμε να του αντικαταστήσουμε, αλλά θα εξηγήσω γιατί τα έχουμε βάλει αυτά τα στοιχεία. Πρώτον, Εάν έχουμε πολύ σημαντικό κλενδυνισμό ανεργίας, αυτό μεταφέρεται με τον καιρό, μετατρέπεται σε μακροχρόνια ανεργία τα δικά μας καθεστώτα ε, θέλουν να, δεν καλύπτουν ε, τη μακροχρόνια ενεργεία γιατί εκεί υπάρχουν σημαντικές διαφορές ε, μεταξύ των κρατών μελών. Όμως μιλάμε για βραχυπρόθεσμους κλειδονισμούς. Κάποιες φορές αυτό βέβαια μεταφέρεται, μετατρέπεται σε μακροχρόνια ενεργεία. Για παράδειγμα, όταν είχαμε αυτό το πολύ σημαντική κρίση στην Ισπανία το 2008-2009, αρχικά έχουμε πολύ ψηλά σημεία αποζημίωσης και μετά αυτό μειώνεται καθώς ε, αυτή η ανεργία μετατρέπεται σε μακροχρόνια. Το δεύτερο στοιχείο που μας περιορίζει είναι αυτός ο, ο μακροχρόνιος ε, κανόνας εξισορρόπησης. Αν έχουμε ένα αθρηστικό έλλειμμα, τότε πρέπει να συμβάλλει περισσότερο. Παίρνει τα ίδια χρήματα λοιπόν, αλλά πρέπει να συμβάλλει σε μεγαλύτερο βαθμό στο Ευρωπαϊκό Ταμείο. Επομένω, το καθαρό ε, όφελο είναι μικρότερο. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που έχουμε θέσει εμείς. Ε, στις επιλογές 1α ε, και 2α δεν υπάρχει. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Για παράδειγμα, στην Ισπανία ή στις Βαλτικέ ε, χώρε, σε όλες τις προσωμιώσεις μας, μετά τα ωφέλη αρχίζουν και μειώνονται ακριβώς επειδή πρέπει να ε, συμβάλλουν περισσότερο. Αλλά στις χώρες της Βαλτικής αυτό δεν είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί ε, ανέκαψε σύντομα η οικονομία τους. Επομένω όλα πήγαν καλά εκεί. Εφόσον όμως στην Ισπανία η ύφεση, στην Ελλάδα η ύφεση κρατά για πολλά χρόνια, πρέπει να ξεκινήσει η μετατροπή όταν βρίσκονται χώρες ακόμα στην ύφεση και στην κρίση. Σε ό,τι αφορά το μέγεθος ε, και των εισφορών και του συστήματος, θα ήθελα να πω τα εξή. Οι διαφορέ μεταξύ των δικών μας προσωμιώσεων και των δικών τους είναι ότι έχουμε μια περίοδο 14 ετών, 99-2012. Έχουμε λοιπόν και καλέ και κακέ εποχέ. Ενώ ε, η προσωμείωση του ΙΖΑ εστιάζει την προσοχή της περισσότερο ε, στις κακές εποχές, στην κρίση τα τελευταία έξι χρόνια και έτσι απαιτεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Εξαρτάται από το τι περιμένουμε για τα επόμενα έτη. Εάν θέλουμε η μέση τιμή από το 99 το 2012 να είναι η μέση μας τιμή, τότε θα είναι πιο φτηνό. Αν πάρουμε μόνο τα χρόνια της κρίσης, τότε βεβαίως ε, το σύστημα γίνεται πιο ακριβό. Το τρίτο σημείο ε, για το χρονοδιάγραμμα το χρονικό, τη χρονική διάσταση. Πρώτον, πόσο γρήγορα μπορεί να ξεκινήσει αυτό το σύστημα. Το εναρμοσμένο σύστημα ξεκινά ελαφρά πιο γρήγορα. Γιατί αυξάνεται ο αριθμός των ανέργων, Επομένω, το Ταμείο αρχίζει και ε, αυξάνεται τις πληρωμές προς ε, την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει λοιπόν καθυστέρηση στο εναρμονισμένο σύστημα. Στο σύστημα καταστροφών η καθυστέρηση εξαρτάται από το στοιχείο της ενεργείας που θα εξετάσουμε. Αν θέλουμε να περιμένουμε τον, ε, τον ετήσιο συντελεστή ενεργείας, θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να βγουν τα στοιχεία. Αν εξετάσουμε τα τριμηνιαία στοιχεία, απαντάμε και αντιδρούμε τρεις μήνες μετά. Αλλά και τα στοιχεία της ανεργίας συνήθω είναι ε, διαθέσιμα πολύ γρήγορα, εντός δύο μηνών από το τέλος περίοδου. Επομένω, η έναρξη λειτουργίας του συστήματος δεν είναι προβληματική. Σε ό,τι αφορά τον χρόνο αντίδρασης λοιπόν και τα δύο συστήματα έχουν ε, ε, σχεδιαστεί με γνώμονα την γρήγορη αντίδραση. Εδώ έχουμε μια διαφορά ε, σε σχέση με το αμερικανικό σύστημα. Εκεί Υπάρχει ε, πολύ ε, μεγάλος βαθμός ισορροπίας μεταξύ των πολιτιών. Όταν βρίσκεται μια πολιτεία σε έλλειμμα, πολύ, πολύ γρήγορα πρέπει να περάσει σε εισφορά, σε μεγαλύτερη εισφορά. Όμως, κάθε φορά που υπάρχει η ύφεση, το Κογκρέσο παίρνει και έκτακτα μέτρα πέραν των ε, συστημάτων τους. Πέραν λοιπόν του βασικού μηχανισμού μπορούν να πάρουν και άλλα έκτακτα μέτρα. Και πάλι είναι πολιτική απόφαση. Όμω δεν θεωρούμε ότι στην περίπτωση Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή σε περίπτωση κρίση εντό ενό μηνό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Επιτροπή να ε, συμφωνήσουν. Γι' αυτό θέλουμε να αποφασίσαμε να το εξετάσουμε με αυτόματο μηχανισμό. Κάτι το οποίο είναι πιο κατάλληλο για τις ευρωπαϊκές δομές διακυβέρνησης. Τώρα για το πόσο γρήγορα μπορεί να συσταθεί ένα τέτοιο μηχανισμός, Πρόκειται κατά κύριο λόγο ε, για νομοθετικό και πολιτικό ζήτημα. Στην εφαρμογή του είναι εύκολο και απλό και γρήγορο. Χρειάζεται όμως γρήγορη μεταφορά σε ό,τι αφορά το ενεργομένο σύστημα. Στην περίπτωση των καταστροφικών αποζημιώσεων δεν χρειάζεται καν μεταφορά. Γιατί πρόκειται μόνο για χρηματοοικονομικές μεταφορές ε, μεταξύ ευρωπαϊκού και εθνικού συστήματος. Εάν περάσει λοιπόν ο κανονισμός θα μπορούσε να συσταθεί πολύ γρήγορα του χρόνου για παράδειγμα. Δεν υπάρχει περιορισμός εδώ. Το μειονέκτημα του καταστροφικού συστήματος είναι ότι στα αρχικά συστήματα πρέπει να γίνει μία οικοδόμηση, ένα build-up για να διαμορφωθεί το αρχικό αποθεματικό. Τώρα, κατά πόσο είναι κάτι το επίγον για την Ευρώπη, τελευταία μου παρατήρηση, αυτό εξαρτάται ε, από το βαθμό των κλειδονισμών που αναμένουμε στην Ευρώπη τα επόμενα 5-10 χρόνια. Εάν ε, περιμένουμε και αναμένουμε η ευρωπαϊκή οικονομία να μοιάζει περισσότερο με την οικονομία μας το 97-2007, τότε ο κίνδυνος είναι χαμηλός γιατί οι χώρες που θα είχαν αποφεληθεί πριν από την κρίση αφορά μόνο σύντομες περιόδους για τις χώρε τη Βαλτική, μικρές περιόδους ε, για την Ισπανία, αλλά δεν είναι πολύ σημαντικός ε, ο κίνδυνος. Εάν περιμένουμε περίοδος 2007-2012 ε, να είναι κάτι το έκτακτο και ότι δεν θα ξανασυμβεί, τότε δεν είναι πολύ επίγον. Εάν περιμένουμε ότι αυτό, τέτοιοι κλειδονισμοί αντίστοιχη σοβαρότητα θα επανέλθουν, τότε είναι πιο επίγον. Επομένω, εξαρτάται από το... τι προοπτικέ που έχουμε για το μέλλον. Ευχαριστώ. Να προσθέσω ε, μερικά στοιχεία στα όσα είπε ο συνάδελφο. Πρώτον, για τον αντίκτυπο στο... κατά τον πρώτο έτο τη κρίση. Αυτό είναι κάτι που εμείς έχουμε θέσει, ένα δικό μας στοιχείο, όμως δεν ισχύει τόσο στην καταστροφική ασφάλιση. Γιατί έχουμε πει ότι όταν η ανεργία είναι πάνω από ένα βαθμό, ένα ποσοστό, και αυτό μπορούμε να το εξετάσουμε, τότε η χώρα που αντιμετώπιζε πρόβλημα λαμβάνει χρηματοδότηση. Αυτό μπορεί να ξεπερνά τον ένα χρόνο. Δεύτερον, πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για να θεσπιστεί το σύστημα. Μπορεί να γίνει σχετικά γρήγορα, αλλά με διαφορετικές ανάγκες μεταξύ των δύο συστημάτων. Αν πάμε στο αρμονισμένο σύστημα, υπάρχουν σημαντικά διοικητικά εμπόδια. Πολλά στοιχεία θα πρέπει να επιληφθούν διασυνοριακά. Ενώ ε, στην καταστροφική αποζημίωση, ε, δημιουργούμε ένα ταμείο και μεταφέρουμε, διαβιβάζουμε ε, τα ποσά. Επομένω, οι διοικητικέ διαδικασίε είναι πολύ ε, λιγότερε. Um, Να προσθέσω δύο στοιχεία ακόμα για το ποσοστό κάλυψης. Στη δική μου παρουσίαση δεν σας δείχνω το ποσοστό κάλυψη των εθνικών συστημάτων, αλλά του συστήματος Ευρωζώνης. Και αυτό εξαρτάται και από τις ε, πολιτικές παραμέτρους. Θεωρούμε ότι όλοι οι νέοι άνεργοι είναι επιλέξιμοι στην Ευρωζώνη. Και είναι επιλέξιμη για ένα δωδεκάμινο κατά μέγιστο βαθμό. Βεβαίως το ποσοστό κάλυψης εξαρτάται και από τις αλλαγές στο ποσοστό ε, ανεργίας, αλλά και στο μερίδιο της, ε, του ποσοστού ανεργίας, στη συνολική ανεργία. Νομίζω ότι ε, ρωτήσατε ε, για το Λουξεμβούργο. Εκεί υπήρξε μια πολύ σημαντική αύξηση του ποσοστού ανεργίας ε, κατά τα έτη 2012-2013 και γι' αυτό το ποσοστό κάλυψης είναι ε, σχετικά σταθερό ή μάλιστα αυξάνεται ελαφρώ τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο τέλος της ακρόασης, αλλά ήρθε και ο συνάδελφος Σέρκας, δεν ξέρω αν θέλουν και οι να μείνουν ακόμα πέντε λεπτά. Παρακαλώ. Ε, Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους παρουσιαστές διότι μας υπέβαλαν ε, μία μελέτη με πραγματικές ε, προσωμιώσεις αλλά στην πολιτική ζωή δεν ξέρω κατά πόσο οι άνθρωποι διαβάζουν, διαβάζουν το πολύ πολύ περιοδικά, αλλά όχι τέτοια έγγραφα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει μία μακροχρόνια θεώρηση των πραγμάτων. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπορούμε να δίνουμε ε, βραχυπρόθεσμα απαντήσεις. Εν πάση περιπτώσει, παρακολουθούμε τις εξελίξεις με μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ ήμουνα σκεπτικιστής στην αρχή, αλλά αρχίζω και κατανοώ την ε, μεγάλη δυναμική αυτής της ε, στρατηγικής και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ένας ε, οικονομικός αλλά και ε, κοινωνικός εξορθολογισμός αλλά με βάση τον ορθολογισμό της οικονομίας και του ε, κοινωνικού ε, τομέα μπορούμε να συγκλίνουμε. Και το ΕΛΚ δεν το βλέπει ε, ιδεολογικά το ζήτημα. Όλοι βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο, στην ίδια κατάσταση. Εγώ είμαι Ισπανός, δεν ξέρω κατά πόσο βοηθηθήκαμε αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια της ε, κρίσης, αλλά ίσως αύριο να είναι κάποιος άλλος θα ήθελα να ευχαριστήσω για τις παρουσιάσεις και ελπίζω η προσπάθειά σας να ε, μην γίνει εν κενό και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε καταρχήν διαβάζοντας αυτές τις μελέτες. Θα μπορούσα να προτείνω στους εμπειρογνώμονες για δύο λεπτά ο καθένας να μας πούν ε, ποια είναι η προστιθέμενη αξία ενός τέτοιου προγράμματος, ευρωπαϊκού προγράμματος αντιμετώπισης της ανεργίας. Maybe, maybe I start, um... Θα ε, πω λίγα λόγια ε, Η τελευταία κρίση κατέδειξε ότι ορισμένα ε, κράτη που επλήγησαν δεν άφησαν το εθνικό τους ε, σύστημα να λειτουργήσει όπως θα έπρεπε προβάλλοντας έναν αυτόματο μηχανισμό σταθεροποίησης. Αυτό είναι και η προστιθέμενη αξία ενός ε, συγκεντρωτικού συστήματος, δηλαδή σε κεντρικό επίπεδο θα προβλεφθεί ένας μηχανισμός σταθεροποίησης και έχει σημασία να τονίσουμε ότι υπάρχουν και εμπλεκόμενοι κίνδυνοι που θα πρέπει να αποτιμηθούν σωστά. Δηλαδή διοικητική χειραγώγηση, κίνητρα των κυβερνήσεων για να αντιμετωπίσουμε τις ε, διαρθρωτικές αδυναμίες της ε, οικονομίας και ούτω καθεξής. Αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν θέλουμε να δούμε πώς θα ορίσουμε ένα σύστημα σε επίπεδο ευρωζώνης. Δηλαδή, πώς μπορούμε να προγραμματίσουμε ένα σύστημα σε επίπεδο ευρωζώνη σε σχέση με τη μόνιμη επανακατανομή και τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια γενική δήλωση. Πρέπει να δούμε τις ιδιαιτερότητες ενός τέτοιου συστήματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η βασική προστιθέμενη αξία είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα όπου οι χώρες να μπορούν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους, γιατί υπάρχει επιχειρηματικός κύκλος που μπορεί να είναι καλός ή κακός. Βλέπουμε όμως ότι αυτός ο κύκλος δεν έχει σωστό άλληλο συσχετισμό με σχήματα απασχόλησης. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια ασφάλιση μεταξύ χωρών όπου όταν τα πράγματα πάνε καλά ε, σε μια χώρα να μπορεί να γίνει χρηματοδότηση σε μια χώρα που δεν ε, τα καταφέρνει τόσο καλά, γιατί ο κύκλος, ε, η κύκλος είναι και γυρίζει και ε, εκεί ακριβώς ε, έγκυται και η επιλογή. Ως προς επιλογές αυτές, θα ήθελα να μιλήσω όχι ως ακαδημαϊκός, αλλά ως πολιτικός. Η βασική επιλογή αφορά τις πιο φιλόδοξες και εναρμονισμένες προτάσεις, οι οποίες θα είναι πιο παρεμβατικές στα εθνικά συστήματα, άρα θα μπορούσαν ε, να ε, είναι πιο δαπανηρά όταν μεταφέρουμε από εθνικό σε ευρωπαϊκό αλλά ίσως υπάρχει μια μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ορατότητα και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα ευρωπαϊκό σύστημα ευημερίας, αν αυτό είναι επιθυμητό τα καταστροφικά, οι καταστροφικές ε, συνέπειες θα ήταν πολύ περιορισμένες, διότι πρέπει κανείς να παρέμβει σε εθνικά συστήματα. Άρα είναι ένα σύστημα που δεν οδηγεί σε κυβερνητικές ε, κρίσεις. αλλά δεν είναι και τόσο φιλόδοξο με βάση την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική. Πέρα λοιπόν από την οικονομική επιλογή είναι και πολιτική. Ποια ε, θεώρηση έχουμε για την Ευρώπη και τι θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό ε, επί του θέματος. Εσείς είσαστε ε, καλύτεροι εμπειρογνώμονες από εμάς. Ναι, πρέπει να χτίσουμε στην προστιθέμενη αξία της δικής σας εργασίας και άλλων. έτσι ώστε να παραμείνουν αυτές οι ιδέες επιτάπητος. Γιατί αν δεν θέλει κανείς την ένωση της μεταφοράς των μεταφορών, σημαίνει ότι θα πρέπει να βρούμε άλλα σχέδια ε, εξισορρόπησης των οικονομικών κύκλων. Χαίρομαι γιατί και εμείς συνεισφέραμε σε αυτή τη συζήτηση. Βεβαίως θα δοθεί περισσότερο input και προσθέμενη αξία, αλλά η δική σας συνεισφορά ήταν πολύ μεγάλη. Ένα πολύ βασικό βήμα. Δεν υπάρχει ομοφωνία επί του θέματος. αλλά χαίρομαι γιατί συνεισφέραμε και εμείς. Και σας ευχαριστώ για, την, για τις πρώτες αυτές μελέτες. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο, αλλά θα επιβεβαιωθεί. Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.